Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Φτάνουμε στο θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται για το Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό στην ε, Μασαλία, 12 ε, με 17 Μαρτίου. έχετε όλοι τις κάρτες σας, αν ναι. πάμε στην Παράγραφο 1, τροπολογία 6, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφο 1, ε, τροπολογία 7, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Τροπολογία 7. Λήξη της ψηφοφορία. 19 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές Φαίνεται να εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Να ελέγξουμε τη 14. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 17 κατά. Ελέγχουμε τη 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18. Συγγνώμη. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19. Σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, επίσης απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 3 αποσύρεται. 4 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και φτάνουμε στην οριστική ε, ψηφοφορία, στην τελική ψηφοφορία, ε, ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 48 υπέρ, κανένας κατά. Καμία αποχή. Θέρμα συγχαρητήρια στους ε, εισηγητές. Στάνουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξη. Ε, την ε, ψηφοφορία για ε, τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικού γιατρικούς σκοπούς. Εδώ είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Ε, ας εργαστούμε λοιπόν όλοι συγκεντρωμένα. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ανακοίνωση. Έχουμε εδώ πέρα μία ε, ψηφοφορία πολλών μαζί. Ε, για κάποια θέματα τα οποία ε, υπάρχουν σε πολλά σημεία του κειμένου. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, αλλά συμφωνήθηκε έτσι με τους κοιόδης εισηγητές. Επίσης, ε, απαράδεκτες έχουν εκριθεί οι εξής τροπολογίες κατόπιν συνεννόησης με την νομική υπηρεσία, οι 240, οι 272, 273, 274 και 275. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η συγγήτρια ζήτησε το λόγο παρακαλώ. Με δώσετε λόγο κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, άκουγα ελληνικά. Κατά λάθο, γι' αυτό δεν σα κατάλαβα. Είχαμε μόνο μία ανταλλαγή απόψεων, ελάχιστη συζήτηση για τις τροπολογίες και λίγα λεπτά για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους και οδησηγητές για την ε, ανεκτήμητη συνεισφορά τους ε, στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Είχαμε 13 συμβαστικέ ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ την κυρία Λόγκ, την κυρία Ζάχου Γκέρλινγκ Γκόρτα και τον κύριο Σλέιτερ, το μοναδικό άντρα σκιώδη συγγητή για την έκθεση αυτή δεν πρόκειται να σας επισημάνω τη σημασία που έχουν τα κείμενα αυτά για τα βρέφτα μικρά παιδιά και για ανθρώπους που χρειάζονται ειδική διατροφή. Τα ενιαία ή συμβαστικά κείμενα μας επιτρέπουν να καλύψουμε το σύνολο των ανησυχιών και των προτεραιοτήτων μας, όπως προέκυψαν από τη συζήτηση, Τώρα, για να είμαι λακωνική, σε ό,τι αφορά το επίμαχο ζήτημα της γλουτένης και της, της ανεξίας στη γλουτένη ή όσοι, τα προβλήματα όσων πάσχουν από κοιλιοκάκι. Είναι πολλοί αυτοί που πάσχουν από κοιλιοκάκι. Δεν είναι μόνο Ιταλοί, γιατί δόθηκε εντύπωση ότι πρόκειται για ένα Ιταλικό λόμπι και μάλιστα η κυρία Σόμερ συμμετείχε στην εκπόνηση της πρότασης, της ενοποιημένης πρότασης, υπαριθμό 5, που είναι απλή και προβλέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το νομικό πλαίσιο να, προ... να προσαρμοστεί σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και την ετικετοθεσία σε αυτό που έχουμε σήμερα. Ούτε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Γιατί αυτό που έχει προταθεί ήταν η επαναχώρηση. Και το επαναλαμβάνω εδώ, γιατί αυτό που έχει το Συμβούλιο επιτάπητο, όπω και η πρόταση τη Επιτροπή που ε, μας παραπέμπει στα health claims, στους χειρισμούς για την υγεία, δεν προστεύει αρκετά όσου πάσχουν από κοιλιοκάκι ή έχουν δυσανεξία στην γλουτένη. Το ενοποιημένο κείμενο επτά αφορά την ετικετοθεσία, την παρουσίαση και την διαφήμιση για προϊόντα όπως είναι παρασκευάσματα για βρέφη. Εκεί προσπαθήσαμε να έχουμε έναν ομοιόμορφο χαρακτήρα και παρόμοια προστασία και για τα δύο. Ε, το ενοποιημένο κείμενο 12 ε, υπάρχει και εδώ το επιμάχο θέμα της απαγόρευσης της διαφήμισης. Έχουμε μια διαφωνία που είναι κλασική και χαρακτηριστική και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας. Η κυρία Σάρμπου επισήμανε το πρόβλημα της Ρουμανίας, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί της. Πάντως είμαι εμ, ικανοποιημένη για την πλειοψηφία όσο ό,τι αφορά την επαγρύπνηση σε όλες τις ε, το σημείο 9 για τα φυτοφάρμακα και για το πακέτο για τα νάνο υλικά. Ένα άλλο θέμα, τα γκάμς. Ε, ε, δεν ξέρω, θα γίνει children's milk, Εμ... Ε, προϊόντα που δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια. Η συμβαστική τροπολογία 6 ανταποκρίνεται και διασκεδάζει όλες τις ανησυχίε, Επί του παρόντος δεν έχει ε, θέση στο πεδίο εφαρμογή, αλλά ζητούμε μία εμπεριστατωμένη έκθεση από την Επιτροπή για το θέμα αυτό. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ε, ξαναδίνω τη σκητάλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίς. Ε, ξεκινάμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Καταρχήν, C1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C2, συμβιβαστική 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C3 υπέρ. Κατά. αποχές. Ας την ελέγξουμε αυτήν, την C3, την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. C4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. C6. Σας παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ, να σηκώσει το χέρι του. Ωραία. Κατά αποχές εγκρίνεται. C7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συ 10 υπέρ. Συ 10 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συ 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται. Συ 12. Ποιος είναι υπέρ. Να ελέγξουμε την C11. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στην C12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. C13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε στις ε, στις block votes, ε, στις ε, ψηφοφορίες όπου ψηφίζουμε πολλά θέματα μαζί. 58-60 μέχρι την 149 και κατόπιν τα εκτιμώντας 66 ε, έως 73. Ε, Ποιος μπορεί να συμφωνήσει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Έτσι λοιπόν γλιτώσαμε πάρα πολύ δουλειά. Φτάνουμε στα επιμέρους άρθρα. Άρθρο 1. Τροπολογία 57 ε, στη σελίδα 15 για μένα. Φτάσατε όλοι στη σελίδα 15. Ποιος είναι υπέρ της 57. 57 υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Δεν είναι σαφή τα πράγματα. Ελέγχουμε την 28. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. Ε, η ΙΜΚΟ 14 είναι η επόμενη την οποία ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 15 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά Αποχέ απορρίπτεται. 133, 133. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Ε, η 30, η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143. Ποιος είναι υπέρ. Να ελέγξουμε την 30. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 33 υπέρ 27 κατά. Ε, ευτυχώς που ελέγξαμε. Ελέγχουμε την 143. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 31. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ σαφές. Ας ελέγξουμε την 31. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το άρθρο 2. Τροπολογία 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Να ελέγξουμε την 146. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 34 κατά. Προχωράμε στην 147 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Dann haben wir zwei identische IMCO 8. Έχουμε δύο όμοιες, την IMCO ε, 34 ε, και την IMCO ε, 18, ποιος είναι υπέρ κατά, εγκρίνεται. Ε, άρθρο 3, 173, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, η 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 179, 181, 19, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρα 17, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 180, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 20 και Ήμκο 21. Να ψηφίσουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συγγνώμη λέει κάποιος. Το 77 δεν έπρεπε να είχε καταπέσει όταν εγκρίναμε την 78. Α, κατάπεσε, οκ. Συνεχίζουμε. 38 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 14 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 και 184 είναι όμοιες τη ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 185, ε, διορθώνει ο πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 192 Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 34 κατά. Απορρίπτεται. 189 υπέρ, κατά, απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 196 υπέρ, Ψηφίζουμε την 196. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ε, απορρίπτεται. Την 44. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε, διότι δεν είναι τελείως σαφές. Είπε, ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 44. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. Φτάνουμε στην ΙΜΚΟ 24. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209. Ποιος είναι υπέρ? Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 25 υπέρ. Κατέ αποχές εγκρίνεται. Η 214 220, ε, 221 και ήτρε 22. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε αυτές τις τέσσερις τροπολογίες. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε η λήξη της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. τροπολογία 215. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.17 της Ρενάτε Όμερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.18, 2.22, 2.23 και η 23 είναι όμοιες. Ε, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές εγκρίνονται. Κατόπιν έχουμε τις όμοιες 226, 234. Ε, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτονται η 219 και η 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ας τις ελέγξουμε. 219 και ήτρα 21. Τις ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 37 κατά. Dann geht's weiter mit den Abstimmungen 49 und ITRE 49 και ήτρα 25, μαζί οι δύο αυτές. Είναι σχεδόν όμοιες, ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. εγκρίνονται. 238 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 26 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρα 24 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε κατόπιν την ε, ε απαράδεκτη τροπολογία. Τροπολογία 50 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. 242 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ, κατά, ε, ε, εγκρίνεται. 245 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 246. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ζητείτε έλεγχος. Ελέγχουμε λοιπόν την 246. Αλλά abgestimmt. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος. 247. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προχωράμε με την 253 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Κατόπιν έχουμε την τροπολογία 51, χωριστή ψηφοφορία. Πρώτα θα ψηφίσουμε το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές. Να την ελέγξουμε. Ελέγχουμε το πρώτο μέρος της τροπολογίας 51. Ah, Λήξη της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 37 κατά. Μόλις με ενημερώνουν όμως δεν προσέξαμε. Το πρώτο μέρος καταπίπτει. Το δεύτερο μέρος όμως πρέπει να το ψηφίσουμε με προφορική τροπολογία. Ε, υπέρ, παρακαλώ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 249, υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 251. Να ελέγξουμε την 250. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 30 κατά, εγκρίνεται. 251. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 253 52 αρχή της ψηφοφορίας. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 252 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 28 κατά. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 259-260 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 261 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 52, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί την 263, την 265 ε, και την 267, ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται με μικρή πλειοψηφία. Ψηφίζουμε μαζί την 53 και την 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε Dann stimmen wir nur ab über 270. Την 270 ψηφίζουμε υπέρ. Ψηφίζουμε την 276 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Προχωράμε στην τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Φτάνουμε στην 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Wir stimmen dann einmal ab über 8. Ψηφίζουμε τις 8 και 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε μαζί τις 10, 11 και 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να την ελέγξουμε. Να ελέγξουμε τη 13. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται η 13. Ψηφίζουμε την 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο Τις 14. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 54 υπέρ, 7 κατά. Ε, ευρία ομοφωνία, αλλά θελήσατε έλεγχο. Ε, οπότε εκπληρώσαμε την επιθυμία σας. Προχωράμε τώρα στην Ήτρε 5. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Η 17 αποσύρθηκε. 84. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 18. Υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Η 36. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 87 και οι 6 θα τις ψηφίσουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 91. Την ψηφίσουμε με προφορική τροπολογία. Παρακαλώ. Είπαμε ότι αν υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική ερώτηση δεν ψηφίζουμε. Αυτό είναι ο κανόνα. Εγώ είμαι κατά τη προφορική ερώτηση. Πολύ χαρίσω ψηφίσουμε την τροπολογία μόνο. Είμαι κατά τη προφορική τροπολογία. Εντάξει, ακούσαμε αντίρρηση ω προ την προφορική τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Ποιο είναι υπέρ του αρχικού κειμένου τη τροπολογία 91. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 πρέπει και εδώ να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 104. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 29 κατά. Με καμία αποχή εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 και 108 ε, της ηγητρίας ε, ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. Προχωράμε κάποιες σελίδες. Επόμενη τροπολογία είναι η 27. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 και ΙΜΚΟ 13 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε. Την 119 και την Ήτρα 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, κάποιος επιθυμεί έλεγχο της 119 και της 11. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. Αυτό δεν φαινόταν από εδώ. 120 και ήτρε 12. Υπέρ είναι όμοιες. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου έκθεση Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε αρχή τη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. 61 υπέρ. Κανεί κατά. Καμία αποχή. Ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε και όσον αφορά το σχέδιο νομοθετικής έκθεση. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσαμε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 62 υπέρ. Καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στη συνάδελφο Ορίστε τι γίνεται όταν οι γυναίκες ασχολούνται αποκλειστικά με έναν φάκελο. Ε, μπράβο σας. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Η συνάδελφος θέλει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ φυσικά να συγχαρώ την εισηγητριά μα, Αλλά α μην ξεχνάμε και του υπαλλήλους γραμματεία που ήταν αρμόδιοι για την ψηφοφορία γιατί ήταν πολύ καλά καταρτισμένος ο κατάλογος ψηφοφορία, και χάρη στη σωστή αυτή οργάνωση από τη γραμματεία καταφέραμε να διεκπαιρεώσουμε εύρυθμα μια αρκετά δύσκολη ψηφοφορία. Θερμά ευχαριστώ λοιπόν και προ τη γραμματεία. Πολύ σωστή παρατήρηση. τι γυναίκες ε, ευχαρίστησα, συμπεριλαμβανομένης ε, και της υπεύθυνη από τη Γραμματεία. Φτάνουμε τώρα στην έκθεση Λάινεν. Σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη. Αναθεώρηση του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Καταρχήν, έχουμε την τροπολογία. Σας παρακαλώ, στην ενδιαφέροντα μπορούν να καταλήψουν την αίθουσα. Και σας παρακαλώ ήσυχα για να ξεκινήσουμε εμείς με την τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε. Να ελέγξουμε την τροπολογία 14. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 27 κατά. Εγώ παραλίγο να έλεγα ότι είναι, εγκρίνεται σαφώς. Ε, τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 έχει αποσυρθεί, 28 της Όσα Westlund υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ήταν σαφές. Προχωράμε. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να την ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 34. 34. Έλεγχο θέλετε για την 33 ή για την 34. Ωραία, πάμε πίσω. Θα ψηφίσουμε την 33 ηλεκτρονικά, διότι εκφράστηκε τέτοια επιθυμία. 33. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 37 ε, ε, υπέρ, 23 κατά. Ε, πάντως ήταν σαφές. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, το εκτιμώντας σε 10 νέο υπέρ. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται το εκτιμώντας C. Ε, ε, θέλουμε έλεγχο για το εκτιμώντας CD νέο. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 35 κατά. Ήτρε 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σαράντα σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 46 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε με την 47 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53. Πάλι έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Πάλι έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129 της Όσα Βέστλουντ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 76 με προφορική τροπολογία. Αν συμφωνείτε, είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας. Τότε θα ψηφίσουμε την αρχική τροπολογία μόνο, χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της αρχικής τροπολογίας, παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 7. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, έλεγχο θέλουν, θέλει κάποιος. Ελέγχουμε λοιπόν την ενοποιημένη τροπολογία 7. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 95 υπέρ. Ψηφίζουμε την 95. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Weiter mit 107 mit einem mündlichen 107 προφορική τροπολογία. Ποιο μπορεί να συμφωνήσει με την 107 με την προφορική τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 την ελέγχουμε. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Σνέλχαρτ. Προχωράμε στην 120. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία έχουμε του Ντάν Γιόρκενσεν 123 το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130. Χωριστή ψηφοφορία πάλι. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131. Θέλουμε έλεγχο. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 ε, θέλουμε έλεγχο, ακούω. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε η λήξη της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 29 κατά. Το έμπειρο μάτι ζήτησε έλεγχο. Μικρή πλειοψηφία υπέρ. Ενοποιημένη τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την ενοποιημένη τροπολογία 10. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορία. 31 ψηφί υπέρ, 28 κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Προχωράμε με την Ρέγγι 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 13. Ε, επιθυμεί κάποιο έλεγχο για την 148. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 31 ψήφοι κατά. 2-2. Ήτρε 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φτάνουμε στην συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό. Πάμε τώρα στην ενοποιημένη 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την ενοποιημένη 12. Ποιος είναι υπέρ. Α, ε, συγγνώμη, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 29 κατά. Τρία δύο. Συμβαστική 13. Ποιο είναι υπέρ. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 4. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 164. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 11 σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Ήτρε 11 το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε το δεύτερο μέρος της Ήτρε 11. Λήξη της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 24 κατά. Ήτρε 14. Αρχή, ε, χωριστή ψηφοφορία, ε, ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 6 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8. Χωριστή ψηφοφορία το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές επίσης εγκρίνεται. Να διορθώσω. Ψηφίσαμε την προφορική τροπολογία Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος της ε, 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 με προφορική τροπολογία των πρασίνων. Ψηφίζουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος καταπίπτει. Προχωράμε στην 12. Η χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε στην τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ε, σχεδόν τελειώσαμε. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 50 υπέρ, 8 κατά, μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια, Γιώ Λάινεν. Αυτές ήταν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για την επιθαρχημένη εργασία σας. Ήταν ε, αρκετά πολύπλοκες οι ψηφοφορίες μας. Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. So, ich bitte diejenigen, die weiter... Παρακαλώ, όσους θέλουν να παραμείνουν να πάρουν τις θέσεις τους και όσοι θέλουν να καταλήξουν την αίθουσα να το κάνουν ήσυχα ε, ώστε να μην ε, μας εμποδίζουν στι εργασίες μας. Ε, φτάνουμε στο σημείο 12 της ημερησίας διάταξης, προφορική ερώτηση ε, σχετικά με το Ρίο συνήκωση. Ε, δίνω το λόγο στην Κομισιόν, τη Μολακέλα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Okay, thank you, Mr. Chair. Uh, let me... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία ε, για μια σύντομη ενημέρωση για το πού βρίσκεται η προετοιμασία ε, για την διάσκεψη του ΟΗΕ για την ανάπτυξη. Καταρχήν τα πράγματα έχουν αρχίσει να κινούνται πολύ γρήγορα. Τώρα, τέσσερις μήνες πριν από την ε, ε, διάσκεψη. Καταρχήν Είχαμε, είχε ζητηθεί από τις χώρες να δώσουν ε, τις συμβολές τους μέχρι τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα κείμενο διαπραγμάτευσης, το οποίο εκδόθη στο, τον Ιανουάριο και αποκαλείται σχέδιο 0. Θα είναι δηλαδή τα πορίσματα του Ρίο και έπειτα θα αποτελέσει τελικά το αποτέλεσμα που θα διαπραγματευτούμε βγαίνοντα από το Ρίο. από το Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το σχέδιο μηδέν έγινε, έγινε δεκτή σχετικά θετικά και πιο συγκεκριμένα αναγνωρίζεται ότι η πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της άμβλησης της στόχες παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την απόδοση στην βιώσιμη ανάπτυξη. Και άλλα θέματα είναι επίσης ε, υπό εξέταση σε αυτό το έγγραφο, αλλά το έγγραφο διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή δεν εστιάζεται, δεν είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν είναι πολύ λειτουργικό. Πολύ δουλειά ακόμα πρέπει να γίνει ώστε να έχει καταστεί λειτουργικό. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στην αρχή Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη και έπειτα σε... Ε, συνεχίστηκαν εκεί το Φεβρουάριο. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπτύσσει την επόμενη, τις επόμενες του θέσεις οι οποίες θα οριστικοποιηθούν στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 9 Μαρτίου πράγμα που θα είναι ακόμα ένα βήμα μπροστά για την ε, τον καθορισμό των ευρωπαϊκών θέσεων και τον διάσκεψης κορυφής, γιατί και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο πορίσματά του το Ρίο. Οι πραγματικές διαπραγματεύσεις για το Ρίο μάλλον θα ξεκινήσουν μετά από την πρώτη ανάγνωση στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Αρκετά αργά και μετά αυτό θα οδηγήσει σε τελικέ διαπραγματεύσει πριν από την διάσκεψη την ίδια. Να τονίσω κάποια ζητήματα τα οποία διακυβεύονται και για τα οποία διαπραγματευόμαστε. Καταρχήν, επί, επί τη βάση μιας πρότασης ε, αρχικής πρωτοβουλίας της Κολομβίας και της Γουατεμάλα, υπάρχει ε, μια συζήτηση για το κατά πόσο το, και σε ποιο βαθμό το ορίο θα πρέπει να συμφωνήσει επί ή να ξεκινήσει μια διαδικασία για την ανάπτυξη αυτών που αποκαλούνται παγκόσμιοι στόχοι ή στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ώστε να ηγηθούν των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για να, έχουμε, να επιτευχθεί η βιωσιμότητα. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα καταλήξει, αλλά φαίνεται να υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη για το ότι το Ρίο θα πρέπει να καταλήξει σε κάποιο είδους στόχους για να δείξει το δρόμο μετά το Ρίο, για το τι θα πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μετά το Ρίο. Ε, στην στοχοθέτηση αυτή τη στιγμή η Κομισιόν εστιάζει σε ε, κάποιους τομείς όπου θα θέλαμε να εστιαστεί η προσοχή, πέρα από δηλαδή την ε, στοχοθέτηση και την ανάλυση των στόχων της χιλιετίας. Οι πέντε φυτομείς αφορούν τους ωκεανούς, ιδιαίτερα τα αλληλευτικά αποθέματα, την υποβάθμιση της γης, την επάρκεια στο νερό, πέρα από την πρόσβαση στο νερό, που είναι τμήμα της ε, παγκόσμιας στοχοθέτησης, έπειτα χειρισμός των, αποβλήτων, των χημικών αποβλήτων και έπειτα ενέργεια και πρόσβαση στην, ανανε, στην ε, ανανεώσιμη ενέργεια. μετά από τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει ο Γενικός Γραμματέας για την ενέργεια για όλους. Αυτά ήθελα καταρχήν να τονίσω, γιατί είναι αυτά τα ζητήματα που διακυβεύονται. Έπειτα, ένα νέο θέμα έχει ανακοινηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορείς να εξασφαλίσει κανείς ότι οποιαδήποτε στοχοθέτηση να γίνει θα σημάνει εφαρμογή αυτής και εφαρμογή μέτρων ε, ε, σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς για να, επιτευχθεί, να επιταχυνθεί η διαδικασία επιτευχής των στόχων αυτός. Και αυτή θα οδηγήσει ή μήπως θα οδηγήσει μόνο σε οδικούς χάρτες δράσεις. Υπάρχει πολλή δρόμο που πρέπει να διανύσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε πως αυτά τα που θα συμφωνηθούν, ειδικοί χάρτες μάλλον του Ρίου θα είναι επιχείρηση εκεί λειτουργική και αρκετά φιλόδοξη χάρτες ώστε να μπορέσουμε μετά να επιτύχουμε τα όσα συμφωνήσουμε. Τρίτο σημείο είναι το θέμα της διακυβέρνησης. Υπάρχει γενικά συμφωνία για το τωρίο θα πρέπει να συζητήσει τη μεταρρύθμιση μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης βιώσιμης ανάπτυξης. Και βέβαια όλα αυτά συνδέονται με την στοχοθέτηση που θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε θεσμούς που θα αποδώσουν, που θα έχουν επιτυχίες σε αυτά που θα συμφωνηθούν. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι ο περιβαλλοντικός πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυβέρνησης αυτής είναι αδύναμος και κατακαιρματισμένος και γι' αυτό το λόγο το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε ένα θεσμό του ΟΗΕ Υπάρχει ευρύτερη συζήτηση για το, σε ευρύτερες ε, διαπραγματεύσει περί βιωσιμότητα και περί βιώσιμη διακυβέρνησης και με σχετικέ μεταρρυθμίσεις. Τι θα πρέπει να κάνει κανείς για το ΕΚΟΣΕΚ, θα πρέπει να φτιαχτεί ένα νέο συμβούλιο για την βιώσιμη ανάπτυξη από την ε, προοπτική της Ένωσης η συζήτηση θεσμικής μεταρρύθμισης είναι ευρύτερη από ότι ε, απλά τα σώματα του ΟΗΕ. Οι διεθνείς σηματοπιστικοί οργανισμοί και το καθεστώς παγκοσμίου εμπορίου θα πρέπει επίσης να δώσει προτεραιότητα, σύμφωνα με την άποψη της Ένωσης, στις νέες αλλαγές που θα χρειαστούν καθώς και να μεταρρυθμιστεί η συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχει μετακινηθεί από το τοπικό σε τοπικό επίπεδο σε επίπεδο μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και αυτό βέβαια πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Επίσης τελική συζήτηση θα αφορά το μέσα για την εφαρμογή. Ποιος θα πληρώσει τι και για ποιον αν συμφωνηθεί κάτι στο Ρίο έχει αξιολογήσει ότι η μεταρρύθμιση σε πιο πράσινη και πιο ε, ολοκληρωμένη πολιτική θα απαιτούσε ένα ένα 2% ε, επενδύσεις ε, σε σχέση με το ΑΕΠ ετησίως. Και είναι σαφέ ότι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, καμία επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε τέτοια κόστη, ιδιαίτερα στι αναπτυσσόμενε χώρε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καλυφθούν τα δαπάνε αυτέ εθνικά, γιατί είναι προ το συμφέρον κάθε χώρα να δουλέψει για αυτήν την μεταμόρφωση. Και έπειτα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καταλύτες ώστε να κινητοποιηθεί περισσότερο, περισσότερα κονδύλια. Οι απόψεις διαφόρων χωρών και ομάδων χωρών αναπεριφέρει ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σας πω ότι περισσότεροι δέχονται την ιδέα μιας πιο πράσινης και πιο ολοκληρωμένης οικονομίας ως ένα νέο όχημα, μια νέα ευκαιρία ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη που θα παρέχει οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης ταυτόχρονα σεβόμενη τα όρια της ανάπτυξης και δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει δηλαδή ένα νέο, μια νέα και ευρύτερη κατανόηση για όλα αυτά, κυρίως για τα αφρικανικές, από τις αφρικανικές χώρες, αλλά και από χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και κάποιες από τις λατινοαμερικάνικες χώρες όπως το Μεξικό, η Χιλή, η Γουατεμάλα, που κατανοούν πως ε, πρόκειται για κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα, υπάρχει αντίσταση στην πιο πράσινη και πιο ολοκληρωμένη οικονομία σε κάποιες λατινοαμερικανικές χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Βολιβία και η Βραζιλία σε κάποιο βαθμό που δεν είναι ακόμα πεπισμένη ότι είναι σημαντική για την παγκόσμια οικονομία και για το μέλλον. Θέλουν να μάθουν περισσότερα. Η Ινδία επίσης ε, ότι αυτό δεν θα αντικαταστήσει την βιώσιμη ανάπτυξη και ότι θα καλύψει όλες τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης ε, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών αυτής. Και έπειτα υπάρχουν κάποιες φωνές που φοβούνται ότι πρόκειται για ένα είδος διακοσμητικής απόπειρας που κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες. Όπω σα είπα ωστόσο, τα πράγματα τώρα κινούνται πιο γρήγορα και θα επιταχυνθούν προς τον τέλειο Απριλίου-Μάιο στις τελικές διαπραγματεύσει, αλλά ο δρόμος για την εξασφάλιση φιλόδοξιων και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από το Ρίο δεν θα είναι εύκολος. Θα υπάρξει πολύ εσωτερική δουλειά εδώ στην Ένωση, αλλά και ιδιαίτερα εκτός εξωτερική διπλωματία που χρειάζεται για να βρούμε ε, συμφωνίες στο Ρίο που να είναι ικανοποιητικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έπειτα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να παίξουν και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι και η κυρία Καμσκάτε από την ε, Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Θέλετε να πάρετε και εσείς το λόγο. Ε, από ό,τι βλέπω όχι. έχει λοιπόν το λόγο ο συνάδελφος Γεμπράντη. Παρακαλώ. Ενημερώνω ότι και το Συμβούλιο είναι παρόν. Να δώσω πρώτα το λόγο στο Συμβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζω αυτά που ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να υποβάλω και εγώ κάποια σχόλια. Καταρχήν, τι γίνεται με τη διαδικασία Ρίο συν 20. Το Συμβούλιο συμφωνεί απόλυτα ότι ε, θέλουμε να επιτύχει, να στεφθεί με επιτυχία το Ρίο. Μας πιέζει ο χρόνος. Θέλουμε να περιλάβουμε τους ωκεανούς, ε, τα χημικά, διακυβέρνηση και ποιος, ποιοι θα είναι οι νέοι φορείς. Αναφίβολα, η νέα σκηνή, το νέο σκηνικό των διαπραγματεύσεων δεν είναι το καλύτερο. Θέλουμε να αποφύγουμε ο, τη διπλωματία που δεν έχει καμία σχέση με τη βιώσιμη, την φοροανάπτυξη, ανάπτυξη, διπλωματία τύπου νέα Υόρκη, και θέλουμε να αναβαθμίσουμε και το πολιτικό επίπεδο. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στο Ναϊρόμπι, στο Συμβούλιο του UNAP και βλέπω ότι όλο και περισσότεροι ε, πολιτικοί και χώρες στον κόσμο εμπλέκονται στη διαδικασία του Ρίου συν 20. Οπότε αναβαθμίζεται και η διεθνής διαδικασία σε πολιτικό επίπεδο και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλλει στη δημιουργία πολιτικής όθησης και μέσω των ε, δικτύων που έχετε και μέσω των εθνικών επαφών. Επίσης υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κάποια συνάφεια μεταξύ στόχων και δράσεων και σε κυβερνητικό και σε πολιτικό επίπεδο. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, αλλά σίγουρα η Ιδανική Προεδρία στο Συμβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί, όχι να διαψεύσει προσδοκίες ή να τις χαλαρώσει, αλλά ίσα ίσα να εντείνει τις προσπάθειες της, στην τελική ευθεία πριν το Ρίο. Είμαστε σε απόλυτη συμπνία μαζί σας και ε, μας πιέζει ο χρόνος όπως σας είπα. Γίνεται κούρσα με το ρολόι. Θέλουμε να δώσουμε θετικά μηνύματα και επεξεργαζόμαστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο Περιβάλλοντος την επόμενη εβδομάδα και τον επόμενο μήνα θα έχουμε άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στη Δανία. Αν χρειαστεί προσαρμόσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, δυναμική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Και σε διοικητικό επίπεδο έχουμε συνεχείς επαφές και μάλιστα θα υποβάλουμε τροπολογίες ε, για την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα, στις προτάσεις του ΙΕ για το Ρίο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και έχουμε και συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δίνουμε και εκεί το παρόν και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο και κάθε ευκαιρία και σε υπουργικό επίπεδο και σε διοικητικό επίπεδο για διμερείς επαφές ε, και με άλλους σημαντικούς ε, παράγοντες της παγκόσμιας σκηνής. Η πράσινη οικονομία δεν εξυπηρετεί μόνο τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά θα ωφελήσει και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό και θα πρέπει να το διατρανώσουμε στο μέλλον. Επίσης, θα φροντίσουμε να δημιουργήσουμε συμμαχίες με τους πιο προοδευτικούς και φυσικά με τις αφρικανικές χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, κάτι που ήδη ξεκίνησε με επιτυχία στο Ναϊρόμπι την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, θα φροντίσουμε να συμπράξουμε και με επιχειρήσεις, με την κοινωνία των πολιτών, θα έχουμε και με αυτούς συμμαχίες, γιατί θα είναι σημαντικοί παράγοντες και πριν και μετά τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άρον Χάνσεν από την Προεδρία που μίλησε εκ μέρους του Συμβουλίου. Τώρα θα ξεκινήσουμε ε, συζήτηση ε, των Ευρωβουλευτών. Πρώτα ο συνάδελφος Γερπράντη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και θερμά ευχαριστώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο για την ενημέρωσή τους ό,τι αφορά την πορεία των συζητήσεων εν ώψη του Ριό Συνήκωση. Είναι ενθαρρυντική η σύμπνοια Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και δίνουμε πραγματικά τη μάχη μας απέναντι στο χρόνο ε, για να προτάξουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους μας. Είναι κάπως αποκαρδιωτικό αυτό που αναφέρθηκε για τη δύσκολη μάχη που έχουμε και στον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει βέβαια. Έχουμε πολλές ευκαιρίες όμως, ας μην τις υποτιμούμε. Πολλές ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις γίνονται εκ παραλίλου με το Ρίο και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή και για τα θεσμικά όργανα να σημειώσουν πρόοδο και να προσπαθήσουν αισθητά να βελτιώσουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο της διακυβέρνησης. Έχω λίγες ερωτήσεις. Καταρχήν ε, για το συντονισμό Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Στο Ρίο, για παράδειγμα, Ποιο από τα δύο θεσμικά όργανα θα είναι ο βασικός διαπραγματευτής. Από την εμπειρία μας, από προηγούμενες τέτοιες μεγαλεπίβολες διασκέψεις, το θέμα του ποιος θα είναι ο βασικός διαπραγματευτής είναι πολύ σημαντικό. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Επίσης, τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο Ντέρμπαν γινόταν συνέχεια μια αλλαγή, μία μετατόπιση του βάρους. Δεν υπάρχει η ενότητα που υπήρχε παλιά, ούτε στο G7. Τι, γίνει, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί οι δεσμοί που αναπτύχθηκαν στον Τέρμπαν μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών χρησιμοποιήθηκαν για να να δείξει αυτή την κατάσταση. Το σχέδιο 0 ήταν κάπως απογοητευτικό. Μπορούμε λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο στη διαπραγμάτευση ενισχύοντας α, τις επαφές που κάναμε στον Τέρμπαν και καλλιεργώντας τις περαιτέρω. Τέλος, Μία ερώτηση προς το Συμβούλιο, την Προεδρία. Είπατε ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι το καλύτερο σκηνικό για τις διαπραγματεύσει. γιατί φαίνεται ότι πολλά στοιχεία εμπλέκονται στην, στις διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να γίνει μια αναβάθμιση προς το πολιτικό επίπεδο. Και αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αποδείξουμε ότι για μας το Ρίο Συνήκος είναι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε τα συμπεράσματα της Παρασκευής να είναι στεναρά και έχουμε και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της επόμενης εβδομάδας. Ποιες είναι οι προγνώσεις για τις επόμενες εβδομάδες, τι προβλέψεις κάνετε και πώς πιστεύετε ότι θα αναμειχθούν στη διαδικασία αυτή η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ Φλόρενς και κατόπιν ο Τζο Λάινεν. Παρακαλώ κύριε Φλόρενς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γερκράντη που θέσατε την ερώτηση αυτή. Ε, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Και το σχέδιο εγγράφου δεν είναι και τόσο δεν έχει τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ευτυχώς που η Κομισιόν ε, συνεχίζει να πιέζει, αυτή είναι και η δουλειά της άλλωστε. Ε, όταν βλέπουμε το τι ε, προέρχεται από την ε, Κομισιόν, ε, ακούσαμε πολύ ε, ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά στο έγγραφο αυτό ε, δεν βλέπω πολλά επιχειρήματα μέσα. Νομίζω ότι απέχουμε πολύ από τις πραγματικές επιτυχίες. Και δεν αναγνωρίζω και την πραγματική στρατηγική αυτό το ανέφερε και ο κύριος Σέικερ Πράντι. Υπάρχει γνωμοδότηση των Ποτόρθνικ και ε, Πίμπαλξ, αλλά το Συμβούλιο το κάνει αυτό ή μήπως η Κομισιόν. Και μιλάμε πράγματι για την Κομισιόν ή μιλάμε μόνο για τον Ποτόρθνικ και τον Πίμπαλξ. Ε, θα ήθελα πολύ απάντηση στα δύο αυτά θέματα και μια δεύτερη παρατήρηση. Θα ήμουν ευγνώμων ε, αν η συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά ε, όργανα ε, ε, υπάρξει και στο Ντέρμπαν. Θα ήμουν ευγνώμων ε, αν μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε τις εργασίες. Ευχαριστούμε πολύ η Καλχάνης Φλόρενς, ο Γιώ Λάινεν και κατόπιν η Τζούντιθ Μέρκης. Ναι, Τζο, παρακαλώ. Ε, χαίρομαι που ακούω ότι το Συμβούλιο και το και οι Κομισιόν ε, ασχολούνται με αυτή τη διάσκεψη κορυφή, την παγκόσμια διάσκεψη κορυφή. Ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ηγετικό ο ρόλο τη μετά από την ε, συζήτηση περί βιωσιμότητα που διεξάγεται εδώ και χρόνια και δεκαετίε, πιστεύω ότι έχουμε και κάτι να προσφέρουμε. Ελπίζω ότι η πολιτική αφενός θα μιλήσει με μία φωνή, αυτό ήδη το αναφέραμε, διότι η Κομισιόν και ε, Συμβούλιο έχουν ε, εδώ ένα κοινό εγχείρημα και επίσης ελπίζουμε η πολιτική να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να οικοδομηθούν ε, συμμαχίες, διότι ακούσαμε, ε, υπάρχουν και ε, ότι η πράσινη ε, είναι ένα κόλπο του βορρά. υπάρχουν τέτοιες υποψίες. Το καλύτερο θα ήταν να επιτευθούν ε, ε, ε, συγκεκριμένοι στόχοι στο Ρίο. θα είμαστε σε θέση να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους στα πλαίσια διαφόρων τομέων στο Ρίο. Επίσης, ένα θέμα είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Εμείς έχουμε νομοθεσία περί της ε, περιβαλλοντικής λογοδοσίας, το Environmental Accounting. Εάν ε, θα ήταν θετικό στο ορίο να αποφασίσουμε ε, σχετικά με τη συλλογή παγκοσμίων στοιχείων όσον αφορά την ικανότητα των στοιχείων καθώς και τα όρια αντοχής των οικοσυστημάτων. Και Επίσης, ε, θα ήθελα ε, να αναφερθώ στην συμμετοχή όλων των ε, stakeholders, των ενδιαφερομένων. Στο Ρίο 92 είχαμε την Παγκόσμια Ατζέντα 2020 και, 21 συγγνώμη, και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να θεσπίσουμε ένα νέο θεματολόγιο για τη βιωσιμότητα και να το στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. η Γιούτιτ Μέρκη. Και κατόπιν ο Βιτόριο Πρόντι. Παρακαλώ, Γιούτιτ Μέρκη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον συνάδελφο που υπέβαλε την ερώτηση. Και ευχαριστούμε και το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις απαντήσεις. Διαβάζοντας το ενημερωτικό σημείωμα για το Ρίο ε, λέει πολλά και διάφορα και είναι όλα με αν. Αν το ένα, αν το άλλο, θα μπορούσαμε ίσως, είναι πολύ δυνητικό το κείμενο. Και με ανησυχεί αυτή η αβεβαιότητα, γιατί 3,5 μόλις μήνες μας χωρίζουν από την ε, σημαντική αυτή ημέρα, την ε, διορία αυτή. Και ήδη υπάρχει μία ε, αβεβαιότητα και αφησιμία ως προς τους στόχους. Και αν είμαστε τόσο γενικοί και όριστοι και ε, υποθετικοί τόσο κοντά πριν την συνεδρίαση του Ρίου, τι θα γίνει. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αν θα μπορούσαμε, λέμε όμως, να προαγάγουμε ή αν θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε. Ωραία όλα αυτά, αλλά παρά είναι υποθετικά. Εγώ θέλω απτά αποτελέσματα. Τι γίνεται ως προς τα συγκεκριμένα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά, γιατί δεν προσπαθούμε να τα προβάλλουμε και διεθνώς. Ε, δεν μίλησαν μόνο οι Επίτροποι Ποτότσινικ και Πίπορς γι' αυτό, αλλά και η Επίτροπος Χέντεργκάρτ πέρυσι στην Ήτρε. Είπαν ότι ε, θα δοθεί έμφαση στην ε, αηφόρο ενέργεια για όλους. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, θαυμάσιο θέμα. Το θέμα είναι όμως αν παραλυώσουμε το μήνυμά μας προσθέτοντας όλο και περισσότερα θέματα, το αποτέλεσμα θα είναι απογοτευτικό. Μήπως ήταν καλύτερο να προσπαθήσουμε όλες τις ε, ετικέτες που έχουμε στον κόσμο, γιατί έχουμε ετικέτες στο ΡΙΟ, όλες αυτές τις οικολογικές ετικέτες ε, που έχουν κάποια, κάποιο αντίκτυπο. Αν φτιάξουμε ένα σύστημα για να μπορεί κανείς να βλέπει πού είναι η πηγή, ποιος είναι ο αντίκτυπος, ποιο θα είναι το περιβαλλοντικό κόστος, τι είδου ε, εταιρική συμπεριφορά έφερε το προϊόν στην αγορά και με τη χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο χρήσιμο. Αν αυτή είναι η έκβαση του Ρίο, να έχουμε μία οικολογική ετικέτα που θα στηρίζεται, θα συνδυάζει και το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και να είναι εμφανή όλα αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ καλύτερο. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε μια τέτοια ε, συνολική συμφωνία και για τη διαφάνεια γιατί ουσιαστικά όλοι γι' αυτό ενδιαφέρονται. Την προέλευση των ε, πρώτων υλών και τη συμπεριφορά των εταιριών. Και κάτι άλλο. Το Ρίο δεν θα πρέπει ε, να είναι τελευταία λύση για, τα, για τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί έχουμε σύστημα COP και μακροπρόθεσμη προοπτική για χώρες, για υπήρους, όλα μάκρο δηλαδή, σε μάκρο προοπτική, σε μεγάλη προοπτική. Μέσα μας ενδιαφέρει ο μικρό κόσμος, πώς θα μπορούμε να συμβάλλουμε στην καθημερινότητα κάποιου Αφρικανού με μέτρα για ενεργειακή πολιτική και ενεργειακή αποδοτικότητα. Να φανούν αυτά τα μέτρα σε επίπεδο ε, καθημερινότητα, σε επίπεδο πολίτη. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ε, το καλύτερο σύνθημα και η καλύτερη ετικέτα για την ε, διάσκεψη του Ρίου Ευχαριστώ πολύ ο Βικτόριο Πρόντι και κατόπιν ο Πίτερ Λίζε. Ε, Εγώ πιστεύω πως το Ρίο είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χαθεί. Γιατί το Ρίο του 92 ήταν πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς λόγω της, ε, των, νεολογικών πρόοδων που σημειώθηκαν εκεί όπως η βιοπικιλότητα αν θυμηθούμε, αν θυμηθούμε το θέμα της ε, βιωσιμότητας σε υφόρο ανάπτυξη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ θαραλέοι εδώ γιατί ακριβώς χρειαζόμαστε κάποιες ιδέες και κάποιες θεμελιώδεις επιλογές. Κατά τη γνώμη μου αυτές θα πρέπει να είναι πολύ πιο ξεκάθαρες. για τα όσα λέμε πέρα από το ΑΕΠ, beyond the GDP. Πώς όμως το να ξεπεράσουμε το ΑΕΠ μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να επανεφεύρουμε και να επανατοποθετήσουμε τον πολιτισμό μας. Πράγμα που υποδεικνύει κάποιες βασικές αρχές όπως ε, ο κεντρικός χαρακτήρας του ατόμου και η έννοια του κοινού καλού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και πτυχές ισότητος που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και όπως για παράδειγμα η πρόσβαση στο νερό. για το νερό το πρόβλημα είναι επιλύσιμο από τη στιγμή που έχουμε την ενέργεια. Αλλά όλοι οι άλλοι φυσικοί πόροι, για τις οποίους δεν έχουμε καμιά βάση, καμιά βάση είναι εξωτερική, και άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της ίσης πρόσβασης στις φυσικούς πόρους για τις επόμενες γενναίες. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσουμε να προσδεθούμε σε αυτή την ιδέα ώστε να αποφύγουμε αυτή την κατάληψη της γης και των ε, φυσικών πόρων που είναι από μόνη της κατά της ειρήνης. Θα μπορούσαμε να επιμείνουμε και περισσότερο λοιπόν για την ελληνική και για, γιατί και αυτή είναι ένα βασικό ε, οικοδομικό υλικό για τη συνοχή της κοινωνία μας και για να μπορέσουμε να βρούμε συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά και ευχαριστώ την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τα όσα έχουν κάνει. Δεν μπορώ παρά να τεθώ στη διάθεσή τους ως επίσημος εκπρόσωπος ε, του Κοινοβουλίου στο Ρίο 8 έτσι ώστε να είμαστε... Να, να, να, είμαστε και πιο συγκεκριμένοι για αυτές τις προτάσεις, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να είμαστε πολύ θαραλέοι γιατί πιστεύω πως μόνο έτσι θα μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια πιο βαθιά σχέση τόσο στο επίπεδο των τοπικών ε, κοινοτήτων όσο και στο επίπεδο των διεθνών κοινοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βιτόριο Πρόντι, ο Πέτερ Λίζε και κατόπιν ο Καρλ Σλίτερ. Πέτερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Συμβούλιο και, το... και την Κομισιόν. Δύο συγκεκριμένε παρατηρήσεις από τη δική μου πλευρά. Καταρχήν, υπάρχει το θέμα ε, είναι το θέμα αν θα πρέπει να έχουμε δικό μας οργανισμό ε, περιβάλλοντος ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Ε, έχει αναφερθεί ε, ένα ε, πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Συνεργαζόμαστε στο θέμα αυτό, συνεργαζόμαστε με τον ΠΟΗ, τον Παγκοσμίο Οργανισμό Υγείας. Υπάρχουν προβλήματα στην Παγκοσμία Οργάνωση Υγείας, δεν είναι όλα τέλεια εκεί. Δεν θέλουμε όμως να καταργήσουμε την συνεργασία αυτή. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία. Και ε, το πλεονέκτημα του ΠΟΗ είναι ότι είναι ένας οργανισμός ε, του ΟΗΕ που μπορεί να λάβει αποφάσεις. Ε, συναντώνται οι Υπουργοί Υγείας όλων των χωρών και μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Φυσικά μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά κανένας δεν λέει ότι ότι θέλουν να το καταργήσουν. Ε, για το περιβάλλον δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε συνάντηση των ε, Υπουργών Περιβάλλοντος όλου του κόσμου. Ε, πιστεύω όμως ότι στο περιβάλλον αξίζει ένας τέτοιος οργανισμός. Τα επιχειρήματα κατά είναι ότι δεν ε, λειτουργούν πολύ καλά διάφοροι φορείς του ΟΗΕ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μην έχουμε παγκόσμιο οργανισμό περιβάλλοντος. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν και το Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό και σας παρακαλώ να ε, στηρίξουν τη θέση αυτή που αναφέρεται και στο ψήφισμα. Δεύτερον, ε, με πολύ ενδιαφέρον άκουσα ότι χώρε όπω η Γουατεμάλα είναι υπέρ τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γνωρίζω πολύ καλά τη χώρα, διότι έχω εργαστεί εκεί ω γιατρό και στην ε, χώρα αυτή διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα χάσμα, όπω άλλωστε και σε πολλέ χώρε πολλοί στο μεταξύ έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά στις ε, χώρες ε, αυτές οι υπουργοί δεν συζητάνε μεταξύ τους. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ ΙΠΑ, Κίνας και άλλων. Συμμετείχε και η Γουατεμάλα και είμαι βέβαιος ότι ε, αυτοί που ε, διαπραγματεύονται με την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο πάνω στα θέματα αυτά δεν γνωρίζουν ότι οι Υπουργοί Μεταφορών μας δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Σας παρακαλώ λοιπόν είτε να είμαστε ειλικρινεί ε, και να πούμε ότι είμαστε κατά της βιώσιμη ανάπτυξης ή να πείτε στα Υπουργεία Μεταφορών σας ε, να ε, σταματήσουν να αντιμετωπίζουν έτσι τους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιστεύω πρέπει να το πετύχουμε πριν το Ρίο. Ευχαριστώ πολύ Πέτερ Λίζε, ο Καρλ Σλούτερ, Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για την πράσινη οικονομία. Ακόμα πολύ συχνά τον όρο πράσινη οικονομία, αλλά σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ελπίζω όταν εσεί ε, το αναφέρετε να μην εννοείται ε, οικονομική μεγέθηση με τη βοήθεια τη περιβαλλοντική περιβαλλοντικής τεχνολογίας, αλλά με την ε, ίδιο πληθωρισμό, με οικονομία που θα στηρίζεται στη δανειοδότηση. Δεν είναι πράσινη μόνο από τεχνολογική άποψη οικονομία. Έτσι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μια πραγματικά πράσινη οικονομία είναι αυτή που όχι μόνο είναι ε, αηφόρος από περιβαλλοντική άποψη, αλλά είναι αηφόρος και από παγκόσμια άποψη και από άποψη αλληλεγγύης. Γιατί και οι φτωχότερες ε, χώρες του κόσμου δικαιούνται πιο ακριβωδική κατανομή των ε, πόρων και του παγκόσμιου πλούτου. Αυτό σημαίνει πράσινη οικονομία. Μία λύση που θα στηρίζεται μόνο στην οικονομική ανάπτυξη για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης πολύ συχνά με πρόσβαση, εύκολη πρόσβαση στο κεφάλαιο που δημιουργήσει η οικονομία της φυσαλίδας και σε χρεοκοπίες, σε απότομες οικονομικές κρίσεις και κράχ, δεν θα έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και θα χρησιμοποιήσουμε και πολύ περισσότερους πόρους. Τι εννοείτε εσείς, πώς εκλαμβάνετε εσείς τον όρο πράσινη οικονομία. Ελπίζω να μην εννοείτε μόνο πράσινη οικονομική μεγέθυνση, γιατί είναι ανεπαρκής αυτή η προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Εσείς τι εννοείτε λοιπόν με την πράσινη οικονομία, γιατί για μας η πράσινη οικονομία περιέχει και κοινωνική διάσταση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Μύροσλαβ Όουσκι και μετά η Σαντρίν Μπελία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω το συνειρμό του κυρίου Σλίτερ. Όταν μιλούμε για πράσινη οικονομία στην Ευρώπη, φαίνεται ότι ξέρουμε τι εννοούμε. Όλοι έχουμε συγκεκριμένες απόψεις για το τι σημαίνει πράσινη οικονομία και θα πρέπει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ορίσουμε σαφώς την πράσινη οικονομία. Αλλά για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι δύσκολο να αντιληφθούν ότι η πράσινη οικονομία δεν είναι ένα κόλπο, ένα τέχνασμα των πλούσιων χωρών για να εξασφαλίσουν τη δική τους ανάπτυξη εις βάρος ε, της ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν είναι εύκολο να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω περισσότερες διευκρινήσεις και πιο συγκεκριμένες προτάσεις για την πράσινη οικονομία. Ευχαριστώ τον κύριο Γερμπράντη που υπέβαλε την ερώτηση, τις ερωτήσεις του μάλλον, γιατί χάρη στις ερωτήσεις αυτές μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση παρόλο που έχω και κάποιες ενστάσεις για το secure, για τον όρο εξασφάλιση δηλαδή. Πιστεύω ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο δεν μπορούν να επιτύχουν κάτι σε διεθνές επίπεδο. Μπορούν να δώσουν μια μάχη, να κάνουν μια προσπάθεια, αλλά, αλλά πώς θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταρρύθμιση των ΗΠΑ. Αυτό είναι αδύνατο. Δεν έχει τέτοια δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια εξουσία. Χρειαζόμαστε ε, διεθνή συμφωνία. Μόνο το του οίκου μας εμείς μπορούμε να το μεταρρυθμίσουμε. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεταρρύθμιση σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, το Ρίο Συνήκωση θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο, πιο τοπικό, πιο κοντά στους πολίτες. Συμφωνώ γιατί πολλές φορές προτάσουμε μεγαλεπίβαλους αξιέπαινους βέβαια στόχους και είμαστε υπέρ της αηφόρου ανάπτυξης, αν όμως δεν προτείνουμε συγκεκριμένες αυτές ιδέες, θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ποιε είναι οι πρωτοβουλίε που μπορούν να αξιοποιηθούν και από τι αναπτυσσόμενε χώρε, όπω η διαχείριση των αποβλήτων, η ανακύκλωση των αποβλήτων, καταπολέμηση τη ρήπαση του ύδατο. Νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε και σε αναπτυσσόμενες χώρες κάποιες ευπρόσθετες λύσεις. Και Πηγαίνουμε σε ωραίες χώρες της τροπικής ζώνης, αλλά διαπιστώνουμε με φρική ότι καίνε τα σκουπίδια στις χωματερές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και οι χώρες αυτές να μπουν στον δρόμο της ανάπτυξης, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, αναβαθμίζοντας το βιωτικό τους επίπεδο. Νομίζω ότι τέτοιοι συγκεκριμένοι στόχοι θα τύχουν γενική υποστήριξη, γιατί και στη Μαλαισία και στην Ινδονησία ενδιαφέρονται για την ποιότητα του ύδατό του, για το περιβάλλον του. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο, πολύ ειδικό και που είναι και καταμετρήσιμο και μπορεί εύκολα να ε, υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί πολύ πιο εύκολα από το να απλώς να κουνάμε το λάβαρό μας που θα λέει «Κρυζώστε τη φτώχεια». Δεν μπορεί από μόνη της Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεριζώσει τη φτώχεια σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε κύριε Ούσκη, κυρία Σαντρίν Μπελιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συνοπτική γιατί με κάλυψαν οι συνάδελφοι σε πολλά σημεία. Σημερίζομαι και εγώ την ανησυχία που εκφράστηκε για την αβεβαιότητα και την απροσδιοριστία των στόχων και των δεσμεύσεων γιατί δεν ήταν και πολύ διαφωτιστικά τα σχόλια και απαντήσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής γιατί ποια θα είναι η έκβαση αυτής τη τέταρτη διάσκεψης κορυφή για τη γη. Αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι στη θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής και στην προβολή της θέσης αυτής διεθνώς να έχουμε κάποια μεγαλύτερη σαφήνεια. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Τι έχει έχουμε για έναν ορισμό της πράσινης οικονομίας, της πράσινης ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει όμως και την διάσταση της αλληλεγγύης και της αηφορίας σε έναν μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Σε τι φάση της συζήτησης βρισκόμαστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τόνισε την ανάγκη ορισμού και εχέγγυα αηφόρου ανάπτυξης ε, για το Ρίο που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2012. Επίσης, τι γίνεται σε ό,τι αφορά την πρόταση ε, σύστηση ενός αρεξάρτητου οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Περιβάλλοντος. Τι γίνεται με το καταστατικό, τι προβλέπετε για την αποστολή, τη λειτουργία αυτού του οργανισμού και τον προϋπολογισμό του. Παρακαλώ, σε τι φάση βρίσκονται οι συζητήσεις και για αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε κύριε Μπελία. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο και χρήσιμο το να θέσουμε δηλαδή εδώ κάποια ερωτήματα και να δούμε τι κρύβεται πίσω από τις διάφορες λέξεις, ε, τι καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Όταν εμφανιζόμαστε σε μια τέτοια παγκόσμια διάσκεψη, μήπως θέλουμε να επανεξετάσουμε τις ε, διατυπώσεις μας ε, για να γίνουμε κατανοητοί. Και συχνά υπάρχουν και καθαρά πρακτικά θέματα. Ο συνάδελφος Λίζα αναφέρθηκε στην στο, σύστημα εμπορίας εκπομπών και τις αερομεταφορές. Μπορεί να ε, ακούει κανεί ένα ωραία λόγια, αλλά τελικά ε, τα μέτρα που λαμβάνουν οι διάφορες χώρες θα πρέπει να ανταποκρίνονται ε, στους στόχους αυτούς. και η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τι βαθμό συμμετέχει ε, σε όλη αυτή τη θεματική. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός φορέας σε τι βαθμό συμμετέχει σε αυτά τα θέματα ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν μιλάμε για περιβάλλον, πολιτική, για την αλλαγή του κλίματος κλπ. Ε, έχουμε αναπτύξει ε, μια ευρωπαϊκή διπλωματία κλίματος και περιβάλλοντος, ε, πώς έχει η κατάσταση και όσον αφορά την τη χρηματοδότηση, διότι αυτό είναι τελικά το κρίσιμο ερώτημα στο τέλος κάθε τέτοιας διάσκεψης. Ποιος θα πληρώσει για όλα αυτά. Ε, δεν ε, έχει ξεφύγει αυτό από την προσοχή και των άλλων ε, κρατών μελών. Ποια λοιπόν είναι η στρατηγική όσον αφορά τη χρηματοδότηση από πλευρά τη Κομισιόν και του Συμβουλίου. Μία παράκληση προ την Κομισιόν. Μέχρι τώρα είχαμε την καλή παράδοση η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει απόλυτα, διότι μετά από μια τέτοια διάσκεψη θα πρέπει εδώ στην ε, ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος και σε άλλες ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου να δημιουργήσουμε νομοθεσία. Θα θέλαμε λοιπόν από την αρχή να συμμετέχουμε, να έχουμε συνεχή ενημέρωση όπως την γνωρίζουμε από τις διασκέψεις ΚΟΠ. Στο όνομα της Επιτροπής λοιπόν σας παρακαλώ για κάτι τέτοιο διότι και εμείς θα αντιπροσωπευόμαστε με 11 μέλη στο Ρίο θα είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο να υπάρξει συνένεση ε, για τις ε, θέσεις ε, που θα αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο και σας παρακαλώ λοιπόν η αντιπροσωπεία μας, η αντιπροσωπεία της ΕΝΒΗ από την αρχή μέχρι το τέλος να συμμετέχει στα briefing και όσον αφορά την όλη συνεργασία. Και φυσικά ε, πρόκειται για παράκληση και, τις, και προς την Προεδρία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία. Να δώσω και πάλι το λόγο στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά, ήταν πολύ πλούσια η συζήτηση και όλη αυτή η πληθώρα των σχολείων και των παρατηρήσεων επιβεβαιώνουν την εντύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι υπάρχει σύμπνοια και εστερνιζόμαστε τις ανησυχίες τα δύο θεσμικά όργανα. Ήταν σαφές το μήνυμα από αυτή την άποψη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τώρα στις διάφορες ερωτήσεις. Μας ρωτήσατε πώς θα γίνει η διαπραγμάτευση. Για το αν δηλαδή το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα συνεργαστούν στις διαπραγματεύσεις. Σας διαβεβαιώ ότι η συνεργασία είναι αγαστή, είναι εξαιρετική και έχουμε στενή συνεργασία και επαφές με την Προεδρία και τυπικός και ατύπος και έχουμε συστήσει από κοινού μια διαπραγματευτική ομάδα που παρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από εκπροσώπους αντιπροσωπείας της Εξωτερικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στη Νέα Υόρκη και από εκπροσώπους της Προεδρίας. Σας διαβεβαίω λοιπόν ότι η, η συνεργασία είναι αγαστή και δεν χρειάζεται να αφιέρωνουμε μάλλον χρόνο σε τέτοιε συζητήσει Πάντως και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερωθεί πλήρω στη Νέα Υόρκη. Θα κυκλοφορήσουν και ενημερωτικά σημειώματα, θα γίνονται τακτικά ενημερώσεις και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ ευχαρίστως μάλλον να έχουμε στενή επαφή και με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Νέα Υόρκη. Ένα άλλο θέμα μιλήσετε για τις αναπτυσσόμενες χώρες και το G77. Και αν ε, η διάσπαση του G77 στο Τέρμπαν ε, μπορεί να αξιοποιηθεί από εμά ή αν μπορούμε να βρούμε κάποιους συμμάχους σε ορισμένες χώρες του G77. Βέβαια, η ομάδα των 77 χωρών δεν είναι υπέρ της διάσπασης, δεν θέλει να κατακαιρματιστεί και κάθε πλευρά να πηγαίνει προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά ειδικά οι αφρικανικές χώρες ε, συμπνέουν με την ε, ευρωπαϊκή θέση ως προς το και μάλιστα 62 μέλη της Αφρικανικής Ένωσης ανέκριναν μια κοινή θέση εν ώψη της συνάντησης κορυφής στο Ρίο που είναι πολύ παρόμοια με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έχουμε μόνο τις αφρικανικές χώρες που συμφωνούν μαζί μας. Ακόμη και εντός της ομάδας των 77 υπάρχουν κάποιες διαφορές. Το θέμα είναι ότι ξέρουν ότι όταν έρθουν στις διαπραγματεύσει θέλουν να έχουν συμφωνήσει, να έχουν προσυμφωνήσει σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Κάτι που είναι δύσκολο και αρκετά συντηρητικό από άποψη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνάδελφος Μίκελ από την Δανία όταν μίλησε για διπλωματικές επαφές Νέας Υόρκης και ότι ότι δεν θα πρέπει ε, οι διαπραγματευτές να είναι μόνο διπλωμάτες, εννοούσε ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη για πολιτική ηγεσία στον τομέα αυτό. Γιατί πάλι οι διπλωμάτες, οι διοικητικοί συνήθως δεν είναι θέση να συμβάλλουν σε σημαντική πρόοδο, να κάνουν πραγματικά εντυπωσιακές ε, επιτυχίες. Γι' αυτό και είναι σημαντική η ηγεσία, ο ηγετικό ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήσιμο και ουσιώδης. Το πρωί είπα ότι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο οι δύο επιτροποί Πίμπαλξ και Πατώσινγκ, όλοι οι επιτροποί εμ, συζήτησαν για το Ρίο, για το ποιο θα πρέπει να είναι το πολιτικό μήνυμα του και πώς θα επιταχύνουμε ε, τις διαπραγματεύσεις. Και οι πέντε προτεραιότητες που σας ανέφερα πρωτοστάτησαν και στη συζήτηση αυτή. Θα πρέπει φυσικά να συμβάλλουμε και στο θέμα της επισητιστικής ασφάλειας, αλλά και στο στόχο της εκρίζωσης της φτώχειας. Γιατί αν υποβαθμίσουμε τους φυσικούς πόρους και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτούς, η Χαμένοι είναι κυρίως οι φτωχοί, οι φτωχές χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε και ο στόχος της εκρίζωσης της φτώχειας είναι σημαντικός και δεν θα πρέπει να μεληθεί. Γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια του επιστημιστικού ανεφοδιασμού, που είναι μια άλλη προτεραιότητα του ρίου. Τώρα το σχέδιο 0. Συμφωνούμε ο, μαζί σας ότι είναι κάπως αμφίσιμο, δεν είναι και πολύ συγκεκριμένα, κάπως αόριστο. Είναι μια προσπάθεια το ΟΗΕ να συμπηλήσει περίπου 6.000 σελίδες προτάσεων που δεν είναι και πολύ ομοιόμορφες. Και ακόμη δεν έχει φανεί ένας μύθος κάτι ε, συγκεκριμένο σε αυτό το έγγραφο. Ελπίζουμε να συγκεκριμενοποιηθεί στο μέλλον τις επόμενες εβδομάδες. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης και ενίσχυσης της λογοδοσίας ή τρόπος, κατα... μάλλον, τρόπος καταμέτρησης της πρόοδου. Γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για πρόοδο, δεν μπορούμε να την ποσοτικοποιήσουμε, να την αποτιμήσουμε. Όλα αυτά τα θέματα εξετάζονται πολύ εντατικά. Και σε ορισμένα έχει οριμάσει καλύτερη συζήτηση, άλλα λιγότερο. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να υποβληθούν επιτέλους πιο συγκεκριμένες ιδέες για να έχουμε πιο απτά πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Και τέλος, ορισμός της πράσινης οικονομίας. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να μιλούμε για πράσινη οικονομία που δεν θα αποκλεί κανέναν θα ανοίγει τις αγκάλες της και δεν θα περιθωριοποιεί. Δεν ξεχνούμε λοιπόν και την κοινωνική διάσταση, γι' αυτό και μιλούμε για inclusive economy. Και εμείς ως Ευρωπαίοι με τις πολιτικές μας είμαστε σε καλύτερη θέση για να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Γιατί αν έχει βιώσει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημαντικές επιδόσεις είναι ε, η κοινωνική διάσταση των οικονομικών της πολιτικών. Πάντως, όντως, χρειάζεται σαφήνεια στον ορισμό της πράσινης οικονομίας. Πάντως, θέλουμε ουσιαστικά να προσαρμόσουμε την οικονομική μας ανάπτυξη στην πραγματικότητα που δημιουργούν παγκοσμίως ε, και οι περιορισμοί που υπάρχουν αλλά και οι κοινωνικές ανάγκες. Αυτό θα πει πράσινη οικονομία. Και τέλος, η στρατηγική χρηματοδότησης. Και ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή. Μιλήσαμε για κοινή και αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη και ούτω καθεξής. Εμείς είχαμε στείλει ένα ηχηρό μήνυμα και πολύ σαφές ότι δεν θέλουμε συμπληρωματικούς επίπους αλλά θα πρέπει πρώτα να εστιάσουμε την προσοχή μας στην καλύτερη αξιοποίηση των ε, πόρων. Βέβαια έχουμε την αναπτυξιακή βοήθεια, τις ε, επόμενες χρηματοοικονομικές, ε, δημοσιονομικές προοπτικές, τι γίνεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το μήνυμα πάντως είναι ότι δεν θα αρκέσουν αυτά τα κονδύλια. Ούτε υπάρχει καμία ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει. Είναι και προς δικό μας όφελος όταν μιλούμε για τη μετάβαση ότι είναι προς το περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος της κάθε χώρας να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά όπου χρειάζεται βοήθεια για να έχει κάποιο καταλητικό ρόλο, για να δώσει τεχνογνωσία και συμβουλές για τη δημιουργία δυναμικού, θα δοθεί. Αυτή είναι η χρηματοδοτική μας στρατηγική και γι' αυτό μας ενδιαφέρουν ε, διεθνής ε, χρηματοπιστωτική, ε, μας ενδιαφέρει η διεθνής χρηματοπιστωτική υποστήριξη από διεθνείς φόρες και ατύπως τουλάχιστον υπάρχει συνεννόηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανεπιβεβαιώσει τους στόχους της για το ODA και τουλάχιστον αυτή είναι, αυτό είναι το μήνυμα της δικής μας διεύθυνσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εξασφαλίσουμε και δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς για να δοθούν επενδύσεις και να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δώσω και τον λόγο στο Συμβούλιο, στον Άρον Χάνζεν. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. I'll do this very short. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Και από την πλευρά της Προεδρία θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις και τις, τα σχόλιά σα, τα σημειώσαμε. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω την ανάλυση της Κομισιόν για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσει. Έχουμε εξαιρετική ομάδα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτιάξουμε μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, μια ισχυρή φωνή και φυσικά θα κάνουμε και ό,τι μπορούμε ώστε να συνεργαστούμε μαζί σας, τους ευρωβουλευτές, όταν φτάσουμε στο ε, Ρίο. να αναφερθώ σε μια ερώτηση που, λέ, που ήταν κατά πόσο είμαστε σίγουροι ότι το Συμβούλιο θα στείλει ισχυρά μηνύματα αυτή τη βδομάδα και την επόμενη. Ναι, είμαστε. Είμαστε βέβαιοι πως θα στείλουμε ισχυρά μηνύματα που θα δώσουν κατεύθυνση στη δουλειά μας, στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί οι Υπουργοί Περιβάλλοντος την επόμενη εβδομάδα θα καθορίσουν τις εντολές και θα φτάσουμε πιο κοντά σε έναν ορισμό για την πράσινη οικονομία που δεν θα σας τον αναφέρω τώρα με λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας πω όταν μιλάμε για μια ολοκληρωμένη πράσινη οικονομία για να συμπεριληφθεί εκεί και η κοινωνική διάσταση της πράσινης οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Άρον Χάνσεν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή, τον ε, συνάδελφο Κερπλάντη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Επιτροπή και το Συμβούλιο που απάντησαν σε ερωτήσει μας. Πιστεύω πως έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες, αλλά θα έλεγα ότι όχι ότι λείπει η φιλοδοξία, γιατί έχετε φιλοδοξίες και είστε διαρκώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οπότε μπορείτε καλύτερα να κρίνετε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αλλά επίσης μιλάτε για την ανάγκη πολιτικής ε, ε, που θα πρέπει να παρέμβει. Στο επίπεδο των αρχηγών κρατών σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει επίση δεσμεύσει από πλευρά των αρχικών κρατών. Προσβλέπω λοιπόν στα πορίσματα του επόμενου Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη Παρασκευή. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο όμως, αν θυμηθούμε τον τρόπο που μίλησε το Συμβούλιο για το θέμα της βιοποικιλότητας... και της ε, επάρκειας πόρων, δεν ήταν στο επίπεδο που επιθυμούσαμε για να έχουμε επιτυχές, επιτυχή διάσκεψη Ρίου συνήκωση. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την ευκαιρία που έχουμε στις 20 Ιουνίου και την ανάγκη να φτάσουμε σε, ένα, σε κάποια πολύ ε, ισχύρη διεθνή συμφωνία ή συμπεράσματα. Έπειτα, ακούγοντα τι παρατηρήσει σα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, πιστεύω πω η χώρα ε, υποδοχή, η Βραζιλία, θα μπορούσε να παίξει ρόλο κλειδί. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι ως ευρωβουλευτές για να επηρεάσουμε τη Βραζιλία. Και φυσικά έχουμε τα δικά μας δίκτυα βουλευτών που θα ήταν ίσως πιο πρόθυμα να πιέσουν τις κυβερνήσεις από τις κυβερνήσεις. Έχω εμπιστοσύνη στην διαπραγματευτική ομάδα που έχετε φτιάξει τώρα, Συμβούλιο και Επιτροπή, και είμαι πολύ ευτυχής που έχουμε την Δανική Προεδρία αυτή τη στιγμή αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να φτάσουμε στην πολιτική ηγεσία, γιατί τότε έχουμε περισσότερο, ε, περισσότερα εγώ γύρω από το τραπέζι. Πώς γίνεται λοιπόν να υπάρχει μια συνεπής διαπραγματευτική ομάδα τη στιγμή που οι αρχηγοί κρατών και ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ και θα κλείσω ευχόμενος καλή τύχη και ακόμη περισσότερη φιλοδοξία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Επίσης θα θέλαμε να έχουμε γραπτές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, να ενημερωνόμαστε για την πορεία προς το Ρίο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο που είχαμε αυτήν την συζήτηση. Εντύπωσή μου είναι ότι ε, χρειάζεται σημαντική προετοιμασία και χρειάζεται και ισχυρό μήνυμα, διότι είναι θέμα του αιώνα είναι θέματα που πρέπει να αποφασιστούν και η ευκαιρία που μας δίνεται τώρα όσον αφορά το κλίμα, το περιβάλλον κτλ. θα κλείσει κάποια στιγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες ώστε τον Ιούνιο στο Ρίο να έχουμε μια επιτυχημένη διάσκεψη διότι είχαμε ήδη πολλές διασκέψεις τα τελευταία χρόνια, ενώ και τις διασκέψεις COP. Όταν στην εκλογική μου περιφέρεια μιλάω για διάφορες διασκέψεις, σιγά σιγά βλέπω να σβήνει η πεποίθηση ότι ως Ευρωπαίοι μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αυτές προκλήσεις, ε, πόσο μάλλον με την ε, κρίση που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υποσχεθούμε ένα στον άλλον ότι το επόμενο τρίμηνο θα εργαστούμε σκληρά και θα έχουμε Ε, θα πρέπει να πάμε στο Ρίο και να καταβάλουμε τις καλύτερες προσπάθειές μας ώστε να αποτελέσει επιτυχία η διάσκεψη αυτή, διότι ε, δεν ε, μας παίρνει να έχουμε και άλλες αποτυχημένες διασκέψεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή, ήταν πολύ χρήσιμη και επικοδομητική. Και προσβλέπω στην διάσκεψη ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο επόμενο θέμα, το θέμα υπαριθμών 13. Και Έχουμε και εδώ προφορική ερώτηση της συναδέρφου Μπελιέ. Ε, έχουμε παρούσα και μία ομάδα τηλεοπτική από το τρίτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης και θα ήθελα καταρχήν να να δώσω πρώτα το λόγο στην ε, Σαντρίν Πελιέ για αυτό το καυτό θέμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφής και παιδαγωγική γίνεται. Θα ήθελα και η Επιτροπή Περιβάλλοντος να είναι αρμόδιο όπως η επιτροπές ίντα και ε, ήτρε να κληθούμε να δώσουμε γνωμοδότηση για την εφαρμογή της συνθήκης ΑΚΤΑ, της συνθήκης για την καταπολέμηση παραποίηση και απομίμησης στη γεωργία και στη βιοπικιλότητα. Η ΑΚΤΑ είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα εδώ και μερικές εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν και πολύ επίκαιρο θέμα για 7 εβδομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλούμε συνεχώς για την επίπτωση της συνθήκης αυτής στη χρήση του ίντερνετ και για την πιθανή ασυμβατότητά της με την διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά φαίνεται από την σύνταξη του κειμένου της συνθήκης Άκτα ότι εκτός ότι προσπαθεί να ρυθμίσει την απομίμηση ε, κάποιων αγαθών και ε, την πειρατεία στο ίντερνετ ε, υιοθετεί μια πολύ διασταλτική ερμηνεία σε ό,τι αφορά την ε, ρύθμιση ε, και του προϊόντος του αγαθού που υπάγεται σε προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Και σε αυτό το πλαίσιο έθεσα την ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν θέλουμε σε διεθνές επίπεδο να θεσπίσουμε ρυθμίσεις και να προστατεύσουμε όσοι επιδέχονται διπλώμα των ευρεσιτεχνίας, αυτό μπορεί να ισχύσει για κάποια φάρμακα, αλλά θα καλύψει και τα, τις πορές, κάποια τρόφιμα φυτικής ζωικής προέλευσης, που σήμερα ε, καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εκατοντάδες αιτήματα κάθε χρόνο στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δεν μιλούμε μόνο για γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Έχουμε σήμερα χιλιάδες ε, φυτά και σπόρους που καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ε, δύο μεγάλες πολυεθνικές ζητούν ε, διπλώματα ευρεσιτεχνία, η Μονσάντο και η Σιτζάντα. Θέσαμε το ζήτημα σε νομομαθείς και ρωτήσαμε σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ ενός φυτού ενός είδους ή μιας σποράς που εμπίπτει στην προστασία ενός ε, διπλώματος ευρεσιτεχνίας αλλά εμπίπτει ταυτόχρονα και στην προστασία του κόβε που προσπαθεί να καλύψει ε, την κοινή χρήση αυτών των ε, φυτών ή των, των σπόρων, τι θα γίνει, τι θα επικρατήσει. Οι νομικοί μας είπαν ότι υπερέχει εδώ η προστασία του διπλώματος ευρυστεχνίας, που υπερισχύει του συστήματος προστασίας των πιστοποιητικών των φυτών των σπόρων. Το θέμα της σποράς ε, των σπόρων είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργία του 21ου αιώνα γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η χρήση των αδαφών, η πρόσβαση στην γεωργία και στην επιστηστική ασφάλεια και για πολλούς γεωργούς το θέμα αυτό γύρει και οικονομικά και νομικά εμπόδια γιατί υπάγει την Ευρωπαϊκή Γεωργία στο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φυτών φυτικών και ζωικών προϊόντων. Και στο στάδιο αυτή της συζήτησης, μια και μιλούμε για το γεγονό ότι και η, σπορά, και η σπόρη μας και η γεωργία μας εξαρτάται από την συνθήκη άκτα, θα ήθελα να θέσω μια ξεκάθαρη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη άκτα, ποια μέτρα και ποια εχέγγυα θεσπίζονται ώστε στο μέλλον να εξασφαλίσουμε και την προστασία ε, που υπάρχει ήδη για το πιστοποιητικό ε, φυτικής χορήγησης και την προστασία της βιοπικιλότητας και το μέλλον της ε, πολυμορφίας και της ποικιλομορφίας γεωργίας μας και στα πλαίσια των μέτρων που προβλέπει η συνθήκη άκτα, τι μέτρα θα λάβετε για τους γεωργούς μας και για να εξασφαλίσετε την επισητιστική μας ανεξαρτησία και την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπελιέ. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση ε, Trade. Ο κύριος Πόρης, παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ανέκαθεν της θέσης ότι η Συμφωνία Άκτα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας, στα δικαιώματα δημιουργού, ε, συγγενή δικαιώματα, γεωγραφικές ενδείξεις, ε, ε, εμπορικά σήματα κτλ η άκτα προσπαθεί να καταπολεμήσει την παραποίηση από μίμηση και πειρατεία και στον πραγματικό και στον ψηφιακό κόσμο. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές μας ανταλλαγές με τρίτες χώρες. Αυτό είναι το αντικείμενο της άκτα. Και το γεγονός ότι η Συμφωνία Άκτα καλύπτει όλα τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. είναι συμβατό και ήδη προσδιορίζεται στην Ευρώπη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο από την οδηγία 2004-48 σε ό,τι αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησία και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν ανέκαθεν ε, η ίδια και μάλιστα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κυρία Μπελιέ, την απάντηση στην ερώτηση 147 του 2010 που είχε το ίδιο περίπου περιεχόμενο. Η Συμφωνία Άκτα Προβλέπει όμως και κάποιες εξαιρέσεις για ορισμένα δικαιώματα. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, εκπίπτουν από το τελωνιακό και το ποινικό σκέλος της συμφωνίας και επίσης είναι προαιρετική η κάλυψη για, για το αστικό σκέλος της συμφωνίας. Η άκτα δεν είναι μια συνθήκη που έχει στόχο να καθορίσει την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άκτα δεν προβαίνει σε κανένα ορισμό ούτε του διπλώματο ευρεσιτεχνία, ούτε πρόκειται να επαναπροσδιορίσει τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. Αυτή η συζήτηση είναι τελείως διαφορετική και είναι εύλογο να προστατευθούν από διπλώματα ευρεσιτεχνία ζωντανά ε, φυτά και η άκτα όμως προσδιορίζει κάποιες διαδικασίες νομικές, δικαστικές ή διοικητικές, αστικές, ποινικέ σε ό,τι αφορά το δικαστικό σκέλος και διοικητικέ, σε ό,τι αφορά το ελληνιακο σκέλος και προ... διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η συμφωνία όμως άκτα δεν έχει ως στόχο τον προσδιορισμό του τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Τα συμβαλώμενα μέρη, τα μέρη θα καθορίσουν τους όρους αυτούς. Και τίποτα στην Συμφωνία Άκτα δεν εμποδίζει εξέλιξη μετεξέλιξη αυτών των ενιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η Άκτα προβλέπει και μέτρα εφαρμογής ή συγκαλυμμένα μέτρα εφαρμογής ό,τι αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τους σπόρους. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, η Άκτα προβλέπει κάποια μέτρα μόνο σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία που ήδη υπάρχουν στο ε, νομικό προστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2004. Και μάλιστα η οδηγία 2004 που, το 2004 που σας ανέφερα, που αφορά το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι το νομοθέτημα που μεταφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αστικό σκέλος της ΑΚΤΑ. Το κεφάλαιο αυτό, το αστικό κεφάλαιο της ΑΚΤΑ, είναι το μοναδικό κεφάλαιο, το μοναδικό τμήμα που θα μπορούσε να καλύψει τα διπλώματα τεχνίας. Ευχαριστώ. Σα ε, vielen Dank an die Kommission. Ich habe keine weiteren äh, Σας ευχαριστώ. Εσάς και την Κομισιόν. Δεν έχω κανέναν άλλο στον κατάλογο. Όχι. Θα θέλατε να δευτερολογήσετε κυρία Μπελιέ και να κλείσετε το θέμα. Merci, Monsieur le Président. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ναι, έπρεπε να κλείσω οι ανησυχίες και τα ερωτήματα που με προβληματίζουν εδώ και χρόνια για το μέλλον της ε, βιολογικής ποικιλομορφίας και κυρίως ε, στη Γεωργία. Να σας πω ότι σε σχέση με το άκτα οι απαντήσεις ε, της Κομισιόν αφήνουν ανοιχτά αυτά τα θέματα. Εγώ από ό,τι κατάλαβα οι κυρώσεις της συνθήκης ΑΚΤΑ δεν θα ισχύσουν παρά μόνο στο αστικό δίκαιο, δηλαδή σε ευρεσιτεχνίες. Τι σημαίνει όμως αστικό δίκαιο, αν αύριο μεθαύριο έχουμε μια συγκομιδή βιολογική ή συμβατική καλλιεργία, που κατά λάθο μολύνεται από έναν γενετικό γενετικά τροποποιημένο οργανισμό που εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρεσιτεχνιών. Η αστική εφαρμογή της συνθήκης άκτα θα σήμαινε, γιατί εδώ η, μόλις ήταν, ε, ε, δεν ήταν, ακούσια, τα επέτρεπε στην εταιρεία που έχει στην κατοχή της την ευρεσιτεχνία για το συγκεκριμένο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό να κατασχέσει το σύνολο της παραγωγής. Δηλαδή ο παραγωγός θα στερεί το τις του για εκείνη τη χρονιά. Ξέρετε το πρόβλημα της ε, μόλυσης του μελιού από τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και αυτή τη στιγμή δεν, πριν από κάποιους μήνες και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λύσεις. Δεν έχουμε λοιπόν δυνατότητα εμπορικής αποζημίωσης και δηλαδή αστικής χρήσης του, του άκτα. Το θέμα λοιπόν αυτό ε, υπάρχει και είναι και οικονομικό θέμα και θέμα ελευθερίας για τη γεωργία μας και για τους γεωργούς. Την επιλογή του τι θα ε, καλλιεργήσουν ή θα παράγουν, τι σπόρους θα παράγουν ανάλογα με την επιλογή τους. Θέλει η Κομισιόν να απαντήσει. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Το θέμα της αστικής αποζημίωσης ε, είναι θέμα του δικαστή. Ο θα είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει την, κατά πόσο χρειάζεται αστική αποζημίωση ή όχι. Για να πάρουμε το δικό σας παράδειγμα. Αν είναι τυχαία, η μόλις θα πρέπει να αποδειχτεί ότι υπήρξε βλάβη. Πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές. Πράγμα που δεν είναι σίγουρο. Και ποιος έχει ε, ζημιωθεί αυτός που έχει μολυνθεί ή η η διεθνη ε, πολυεθνική εταιρεία που μιλάει για παραποίηση. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίζουν οι δικαστές, όχι για αυτή η διεθνή συμφωνία. Pour terminer, la Commission euh, répète. Τέλος. Η Κομισιόν επαναλαμβάνει και επιμένει ότι η Συμφωνία Άκτα δεν έχει ως αντικείμενο να ορίσει την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η έννοια της ευρεσιτεχνίας και των πνευματικών δικαιωμάτων, ε, δικαιωμάτων του δημιουργού είναι έγκυρη. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή τη είναι ερωτήματα θεμητά, αλλά τα οποία δεν θα πρέπει να τίθεται σε μια συζήτηση για μέτρα διαδικαστικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας στα ερωτήματα των συναδέλφων και προχωράμε έτσι στο επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη, το υπαριθμόν 14. Έχει να κάνει με τις γεωγραφικές ενδείξεις των αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων. Ο συνάδελφος Παρτολότσι από το ΕΛΚ είναι ο εισηγητής. Του δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση κανονισμού της Κομισιόν, επί τη βάση της οποίας γίνεται η εκθεσή μας, έχει ως στόχο να τροποποιήσει τι μέχρι τούδη ισχύοντα κανονισμό που αφορά την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων, των κοκτέιλ και με βασικό στόχο την βελτίωση της εφαρμοσιμότητας και της αφήνειας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο θέμα. Εισάγοντας μια πολιτική ποιότητα πολύ συγκεκριμένη. Η παρέμβαση της Επιτροπής και ο εξυγχρονισμός ε, τόσο από άποψης ρυθμιστικής όσο και από τεχνικής άποψης έχει οδηγήσει σε, μια, σε κάποιες διατάξεις που μέχρι στιγμής έχουν προστατέψει τον αγορά των αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων που και παρα, και έχουν ε, γίνει σεβαστά από τον γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό στον τομέα των αμπελοϊνικών της Ευρώπης και αποτελούν μια αγορά εξαιρετικά σημαντική από την ποιοτική και ποσοτική άποψη. Ως εισηγητής, συμμερίζομαι τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής και τη γενική προσέγγιση με την οποία γίνεται η προσπάθεια εναρμόνισης του κανονισμού με την ε, νομοθετική εξέλιξη στο θέμα όσον αφορά την πολιτική γεωργίας και όσον αφορά, αυτός όσον αφορά την ενιαία ΚΟΑ, όσον αφορά και τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό το φως των τεχνολογικών καινοτομιών και των νέων προσδοκιών των καταναλωτών. Ταυτόχρονα δέχομαι την, το πνεύμα ευθυγράμμισης ε, του υποεξέταση κανονισμού με τις επιθυμίες των κατανολωτών, τις νέες προσδοκίες των κατανολωτών. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες, 16 ε, τον αριθμό, όπου εξηγούνται οι εξής αρχές. Ευθυγράμμιση του κειμένου και των ε, προσαρτημάτων 1 και 2 με κάποιες ε, τροποποίησεις τεχνικές εκτός από την εισαγωγή των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία των αμπελοϊνικών αρωματισμένων προϊόντων όπως για παράδειγμα η αρωμα... Η προσθήκη ενδεχόμενη του ηνοπνέυματος οι χρωματισ... χρωστικές ουσίες κτλ. Η Ερχή της αποκλειστικότητας επίσης, όπου δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το δεύτερο προσάρτημα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι ονομασίες προέλευσης μάλλον οι γενικότερες ονομασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έτσι ε, να εγγυηθεί την κατάλληλη ποιότητα στους καταναλωτές. Επίσης προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όταν δεν υπάρχει γεωγραφική ένδειξη, αρωματισμένα προϊόντα να δείχνουν στην ετικέτα το όνομα της ποικιλία σταφυλιού που έχει χρησιμοποιηθεί. Τέλος, να εισαχθεί η δυνατότητα για τα αρωματισμένα αμπελοϊνικά προϊόντα να αναφέρουν τη βιολογική φύση των προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί με άμεση αναφορά στην επόμενη, ε, στον επόμενο κανονισμό για τα βιολογικά ε, κρασιά. Στα προστατήματα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, όπως για το βερμούτ, τροποποιήθηκε παρεμβαίνοντας τον ορισμό του αρωματισμένου ίνου με αυγό ε, στην προσπάθεια να προσαρμοστεί στην ειδική μέθοδο ανάλυσης για τη μέτρηση της χολυστερόλης. Τώρα, αν και συμμεριζόμαστε την προσέγγιση προσαρμογής, στην οποία βασίζεται αυτή η πρόταση, έχω υποβάλει μια τροπολογία που έχει στόχο να απαιτήσει μια τέτοια εξουσία να περιοριστεί σε μια χρονική, συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στις γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, εμπίπτει στους στόχους της πρότασης ο προσδιορισμός των βασικών κριτηρίων για την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων. Η πρόταση πράγματι προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τα αρωματισμένα προϊόντα. Ξημερίζομαι τους στόχους της ε, Κομισιόν και στηρίζω την νομική απέτηση και για τα μεταποιημένα προϊόντα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλήρες πλαίσιο όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι οι γενικές γραμμές που ανέπνευσαν την εργασία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε τώρα στον γύρο των σκιωδών εισηγητών. Ο Μάριο Περιλόπου πρώτος, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 1691 από πλευράς της Κομισιόν συνολικά είναι ικανοποιητική. Και έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε έναν ε, θετικό συμβιβασμό για την ασφάλεια του καταναλωτή και το θεμητό ανταγωνισμό ανάμεσα στους παραγωγούς. Η Κομισιόν έθεσε σωστά το στόχο του να φτάσει στον ορισμό που χρησιμοποιείται και σε σχέση με τις νέες τεχνικές εξελίξεις, γραμμίζοντας ε, την ε, πνευματική ιδιοκτησία όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Με αυτή την οπτική άποψη, αυτό που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ, είναι το άνοιγμα στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρασιών και αρωματισμένων ποτών από προϊόντα προέλευσης εκτός Ένωσης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι, πρόκειται για εξέλιξη των ε, παραγωγικών τεχνικών ώστε να λαμβάνονται υπόψη η εξέλιξη που έχει ήδη γίνει στο τομέα, υπάρξει στον τομέα τα τελευταία 20 χρόνια. Ως προς αυτό εύχομαι το Ευρωκοινοβούλιο να μπορέσει να παρέμβει για να τελειοποιήσει περισσότερο την πρόταση μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ρύθμισης των Ενολογικών Πρακτικών που δεν αφήνονται πλέον στην διακριτικότητα της, κάθε, της εκάστοτε εθνικής αρχής. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο μέσω της προσάρτησης ενός νέου παραρτήματος σε αυτόν τον κανονισμό, όσο και με την παραπομπή στη ρύθμιση του τομέα. Συγχαίρω τον κύριο Παύλο Μπερτολότσι για την πολύ ε, ισορροπημένη του πρόταση αναφέρεται και στη βιολογική παραγωγή για τα προϊόντα με βάση το ίνο. Μάλιστα, τις 8 Φεβρουαρίου ε, εκδόθηκε η πρόταση κανονισμού ε, για τα βιολογικά κρασιά. Ε, για το βερμούτ που αρωματίζεται με αυγό. Διάφοροι εκπρόσωποι του τομέα αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά την αύξηση της χολοστερόλης. Δεν είναι αυτό ε, βέβαια, δεν ισχύει βέβαια για τα αρωματισμένα προϊόντα λόγω του φαινομένου της ε, ζύμωσης. Θα πρέπει να γίνεται λοιπόν μια ανάλυση για τα προϊόντα αυτά, όπως αυτός, η ανάλυση που προβλέπεται από τον κανονισμό 110 του 2010. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα, τα, θα μιλήσω δανέζικα. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την ε, δουλειά που έχει κάνει. Είναι ιδιαίτερα τεχνικό το θέμα αυτό. Γενικά, ο καταναλωτής έχει πάντα δικαίωμα να γνωρίζει από πού προέρχεται ένα προϊόν και τι περιέχει. Και γι' αυτό η τεχνική αυτή επικαιροποίηση των ήδη των ε, κανόνων βοηθούν στην απλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων στα πλαίσια των ε, αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων. Έτσι, απλοποιούνται ε, οι προϋποθέσεις για την στρατηγική της ενιαίας αγοράς. Ε, και μέχρι εδώ συμφωνώ. Αλλά όταν μιλάμε για προσαρμογή των ε, ε, λειτουργιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταλαβαίνω πολύ καλά την πρόταση αυτή. Δεν καταλαβαίνω γιατί αποκλείονται τελείω από το παιχνίδι ε, τα κράτη-μέλη και γιατί πρέπει να υπάρχουν πράξη πράξεις ε, σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής, ε, τους περιορισμούς, γεωγραφικές ενδείξεις για να σα αναφέρω μόνο κάποια από τα πράγματα. Και η Κομισιόν επίση έχει πάρει αρμοδιότητα όσον αφορά τι εκτελεστικές πράξει για την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Εγώ δυστυχώς εδώ βλέπω άλλη μία φορά διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, και περικοπή των ε, αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να πετύχουμε την ίδια ομοιομορφία με προαιρετικές, ε, με εθελοντικές διμερείς συμβάσεις. Δεν είναι δυνατόν ο μόνος τρόπος να είναι ε, να δώσουμε περισσότερες ε, εξουσίες ε, στην Κομισιόν για οτιδήποτε κάνουμε εντός της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των σχεδόν εισηγητών. Έχουμε δύο βουλευτές στον κατάλογο των ομιλητών, την Κρίστα Κλάς και κατόπιν Αγιούζο. Πρώτα η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πράγματι είναι τεχνικό το θέμα. Έχουν, υπάρχουν εδώ πολλά διοικητικά θέματα που ρυθμίζονται. Ε, μιλάμε για ένα βιομηχανικό προϊόν. Ε, από την άλλη, για μένα είναι ευαίσθητο προϊόν, ένα ιδιαίτερο προϊόν, επειδή έχει να κάνει με το κρασί. Και, και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ευαισθησία του τομέα. Και δεν μιλάω εδώ μόνο για ένα βιομηχανικό ποτό, αλλά και την πρόσβαση στην οργάνωση αγοράς ε, του ίνου ε, και με τις γεωγραφικές ε, ενδείξεις έχω πρόβλημα. Ξέρω ότι η Γερμανία έχει δύο γεωγραφικές ενδείξεις. Έχουμε το κρασί της Τουριγγίας, αλλά εγώ θα προτιμούσα στον τομέα αυτών να μην ε, μπούμε στο θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων, διότι οι ενδείξεις αυτές προέρχονται από την κοινή οργάνωση αγοράς. Ε, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην συγκριστούμε με τους κανόνες αυτούς. Η Κομισιόν ε, γράφει στην πρότασή της ε, ότι ναι, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις, στους όρους που χρησιμοποιούμε για το κρασί και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλα προϊόντα. Αλλά τελείωσε αυτόματα ε, μπορούν να ε, ε, μπλεχτούν οι έννοιες και να... Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ζημιωθούν οι καλές ονομασίες κρασιών για ένα, από ένα φτηνό προϊόν. Από την άλλη, ο εισηγητής στην έκθεση του γράφει ότι ε, θα πρέπει να δίδεται ε, το είδος ε, των σταφυλιών. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό, διότι μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο περιέχει είναι το οποίο αποτελεί μείγμα διαφόρων και από ένα τέτοιο ποτό δεν μπορεί κανείς ποτέ να γευθεί ένα συγκεκριμένο από μια συγκεκριμένη ποικιλία σταφυλιών. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν η τροπολογίες 2 και 12 να μην υιοθετηθούν. Όσον αφορά αυτά που είπε η συνάδελφος Ρόσμπαχ για τις πράξεις κατοξιοδότηση, αυτά που είπε με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Υπάρχουν ευαίσθητοι τομείς, ε, τους οποίους δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε με κατοξιοδότηση πράξης. Θέλουμε να έχουμε μια κανονική βασική πράξη που να ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Και δεν μας ε, βοηθάει ε, το να θέσουμε προθεσμία στην Επιτροπή. Θα πρέπει μία για πάντα να λύσουμε ε, το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ την προθεσμία. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με πολύ προσοχή, ώστε να, να μην ανατρέψουμε τις καλές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στον τομέα του ίνου. Πρόκειται για ένα βιομηχανικό προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια σωστή ε, ονομασία και ένδειξη για το προϊόν αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κρίστα. Η συνάδελφος Αγιούζα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την έκθεσή του. Αλλά και η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλή είναι και επίκαιρη ευθυγραμμίζεται με τη συνθήκη τη Λισαβόνα με το κανονισμό ε, για την ετικετοθεσία και τι μπελοϊνικές πρακτικές. Καλή πρόταση, καλή έκθεση και χαίρομαι που περιορίζεται η γενική υποχρέωση ε, προσθήκης αλκοόλ για την παρασκευή τέτοιων αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων. Παρόλο που η Σαγκρία βέβαια θα περάσει σε, από 7 σε 4,5 βαθμούς αλκοόλης. Και όσο αφορά τις ποικιλίε, όπως είπε και η κυρία Κλάς, καλό θα είναι να αναφέρονται οι ποικιλίε ε, που χρησιμοποιήθηκαν, ότι ε, είναι υπερβολικό να αναφέρονται οι ποικιλίε που χρησιμοποιήθηκαν για τα αρωματισμένα προϊόντα, αλλά αυτά τα αρωματισμένα αμπελονικά προϊόντα, από τη στιγμή που έγιναν με ε, ίνους παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται να αναφέρονται όλες οι ποικιλίε. Θα πρέπει πάντως να προσδιοριστεί το νομοθετικό κείμενο, αναφέροντας ότι η προστίκη αλκοόλης θα πρέπει να είναι προαιρετική πρακτική ε, διεύρυνσης ε, του φάσματος των φυσικών προϊόντων. Ε, και αυτό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βερμούτ. Υπέβαλα όμως σχετική τροπολογία. Τέλος. Ε, οι όροι σαγκρία και κλαρέα που είναι δύο χαρακτηριστικά τυπικά προϊόντα, τυπικ... ισπανικές σπεσιαλιτέ, θα πρέπει να τροποποιηθούν γιατί για τις χώρες που δεν είναι παραδοσιακά αυτά τα προϊόντα να αναφέροντας αρωματισμένα αμπελονικά προϊόντα με προσθήκη ίσως αγκρίας και κλαρέα. Ο κανονισμός αυτός πέραν της ονομασίας των γεωγραφικών ενδείξεων καλό θα ήταν να αναφέρεται και η εγγυημένη εθνική τοπική σπεσιαλιτέ είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Γιούζο. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, αν θέλει να πάρει το λόγο. Έχουμε τον αναπληρωτή ε, διευθύντη της ΑΚΡΙ, εδώ τον κύριο Λουκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ε, παρατηρήσει, έχω καταγράψει τις παρατηρήσεις. Εν γέννη πάντως φαίνεται να υπάρχει αρκετά θετική στήριξη σε σχέση με αυτή την πρόταση κανονισμού. Όντως ήταν ώρα πια να αναπροσαρμόσει αυτή την νομοθεσία ε, που χρονολογείται από το 1991 ε, έχουν υπάρξει αλλαγές έκτοτε. Οφείλαμε λοιπόν να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό αυτό. Θα αναφερθώ στις παρατηρήσεις των ε, βουλευτών. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το γεγονός ότι ανεφέρεται τα ονόματα των ποικιλιών ε, του σταφυλιού στα αρωματισμένα ποτά. Ξέρετε ότι στον κανονισμό περίνο υπάρχει μια διάταξη που ε, διέπει ε, την δυνατότητα χρήσης ε, της ποικιλία του σταφυλιού μόνο στα ειδικά κρασιά με ΑΟΠ ή ΙΖΠ ε, ή με συγκεκριμένες σοδιές συγκεκριμένων ειδών σταφυλιού. Πολύ αυστηρή νομοθεσία ισχύει αυτή εδώ. Η Διατάξεις αυτές λοιπόν προέρχονται από τον κανονισμό για την ετικετοθεσία του ίνου. Ε, εδώ όμως πρόκειται μόνο για ορισμένε διατάξεις ε, της Κομισιόν δεν αναφέρονται άλλες διατάξεις και δεν αναφέρεται ούτε η γενική διάταξη που προβλέπεται στον κανονισμό για την ΚΟΑ. Θα ήθελα επίση να αναφέρω μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ξέρετε πως διάφορα ποικιλίε συμπεριλαμβάνουν και ονόματα ε, ειδών σταφυλιού. Ε, το Μοντεπουλτσάνο, για παράδειγμα στην Ιταλία, το Βράγκη στην Γερμανία ή Μπουργουνδία για τη Γαλλία. Αλλά στην περίπτωση του Ίνου πολύ περιορισμένη είναι η δυνατότητα χρήσης ονομάτων που συμπίπτουν με τις ε, προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις. Θα πρέπει λοιπόν να ε, σας ειδοποιήσω και να είστε ενημερωμένοι για τις δυνατότητες χρήσης αυτών των ονομάτων των ε, διαφόρων ποικιλίων σταφυλιού για αυτά τα αρωματισμένα κρασιά. Ε, εδώ και λίγο καιρό υπάρχει μια οριζόντια νομοθεσία για τα τους βιολογικούς ίνους και εν πάση περιπτώσει αυτή ισχύει. Δεν βλέπουμε λοιπόν, θα έλεγα ότι υπάρχει μια άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας περί βιολογικών κρασιών εν γέννη. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική ε, γεωγραφικής προέλευσης, η ονομασία προέλευσης, ε, εδώ στον κανονισμό του 1991 προβλεπόταν μονάχα η ονομασία προέλευσης πριν από τις ε, ατυπικές συμφωνίες, τις TRIPS στα αγγλικά και έπρεπε να ενημερωθεί αυτή η νομοθεσία. Υπάρχουν τέσσερις γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης και αυτές πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύονται ως προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις και έπρεπε επίσης, κατά τη γνώμη της Κομισιόν, με στόχο την αναρμόνιση αυτής της νομοθεσίας, να προβλεφθεί και ένα κεφάλαιο για τα ΑΟΠ και τα ΙΖΠ, ΠΟΠ ή ΠΓΕ όπως για τα γεωργικά προϊόντα και τα ε, τρόφιμα. Θέλουμε λοιπόν καλύτερα να προστατεύσουμε αυτές τις ονομασίες προέλευσης και σε σχέση με τις τρίτες χώρες, οι προϊόντα που προέρχονται από αυτές και στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες και γι' αυτό και έπρεπε για αυτά τα αρωματισμένα κρασιά να έχουμε παρόμοιες διατάξεις όπως αυτές που ισχύουν στον υπόλοιπο αμπελονικό τομέα. Για την ε, Σαγκρία... Η Κομισιόν και την, και την Κλαρέα έχουμε status quo που δεν θέλουμε, δεν έχουμε την πρόθεση να το αλλάξουμε. σε σχέση με τον κανονισμό του 1601. Όλοι γνωρίζουμε τη γενικότερη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τις ε, εν πράξης, το κατά πόσο θα πρέπει να αναθέσουμε κάποιες, να τοποθετήσουμε κάποιες βασικές ε, διατάξεις στο βασικό διατακτικό αυτού του κανονισμού παραμένει. Όμως η δυνατότητα για κατεξουσιοδότηση πράξης επιτρέπει στα θεσμικά όργανα να μπορούν να αντιδρούν πιο γρήγορα για την ενημέρωση κάποιων σημείων πολύ τεχνικής φύσης στην νομοθεσία της Ένωσης. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η μέθοδη ανάλυσης. Η ανάλυσης που προβλέπουμε σε αυτήν την νομοθετική πρόταση, η οποία αναφέρεται άμεσα στην ανάλυση του Διεθνούς Οργανισμού ε, του ε, Ίνου και Σταφυλιού και παραθέτεται εδώ και στην ε, ανάλυση μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τέλος θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. E Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρίως όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν ε, με ε, διάφορες συμβολές. Από τα όσα προέκυψαν νομίζω πως η συζήτηση της επόμενης εβδομάδας θα επιστιαστεί σε κάποια ζητήματα τα οποία ήδη αναφέρθηκαν και από πλευρά μου υπάρχει διάθεση για μεγάλη συζήτηση. Αφορά, θα, φορές, θα αφορά μάλλον τις ε, κατεξοδότηση πράξεις ε, για την Κομισιόν, όμως θα ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω γιατί αυτό προβλέπεται από τη συνθήκη όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιστεύω πως ήταν δύσκολο από πλευρά της, του Κοινοβουλίου να αναλάβει μια ολόκληρη σειρά από αρμοδιότητες που είναι πολύ τεχνικής φύσης και που μπορεί να μην επιτρέψουν την ταχεία παρέμβασή μας σε σχέση με τις εξελίξεις. Εγώ ήθελα να... Η δική μου πρόθεση ήταν να περάσουμε σε κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτές τις αρμοδιότητες, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα για πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό το, την πρόταση, κατά τη διάρκεια της του οποίου χρονικού διαστήματος το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει όλες τις επαληθεύσεις, του ελέγχους, για να καθορίσει τη θέση του για αυτό το θέμα. Το άλλο πρόβλημα είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις και η προστασία αυτών και θα ήθελα να υπογραμμίσω πως πρόκειται για κάτι διαφορετικό από το κρασί. Παίρνουμε τις γενικές γραμμές, αλλά τις προσαρμόζουμε σε αυτό το είδος προϊόντος που είναι διαφορετικό από το κρασί, γιατί είναι αρωματισμένο κρασί και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να συγκριθεί με το κρασί. βασιζόμαστε στα γενικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά μετά διαφοροποιούμαστε. Πιστεύω πως θα μπορούσε να είναι μια σημαντική ευκαιρία για να δώσουμε κίνητρα για περισσότερη και μεγαλύτερη ποιότητα για συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτών. Ωστόσο, πιστεύω και από τις παρεμβάσεις που έγιναν ότι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ξανά που πήραν το λόγο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τα όσα υπόθηκαν απόψε. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε αποσαφήνιση και για συνεργασία για τις μελλοντικές ε, τροπολογίες που θα υποβληθούν να, είμαστε, να συνεργαστούμε ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε αυτό το σημαντικό τομέα καθώς και τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Περτολότση. Θα πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες. 8 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και εδώ στις 25 Απριλίου θα ψηφίσουμε το θέμα εδώ στην Ένβη και ε, τον ε, Ιούλιο στην Ολομέλεια. Έτσι ολοκληρώσαμε σήμερα την ημερήσια διάταξη. Θα τα ξαναπούμε αύριο ακριβώς ε, στις 10 η ώρα. Και θα ασχοληθούμε με το θέμα ε, τον, ε, της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στην Ευρώπη. Καλό σας βράδυ.